Mes chers collègues, nous allons commencer. Veuillez prendre place. Συνάδελφοι, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καθίστε. Πάμε λοιπόν. Να ρίξει την καλημέρα, λέει πρόεδρο. Τι κάνει, τι γίνεται, όλα καλά, οικογένεια. Alors, nous ouvrons notre session. Ξεκινάμε λοιπόν στη συνεδρίασή μας. Έχουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξη που αν δεν έχετε αντιρρήσεις εγκρίνουμε ευθύ εξ αρχής. Σημείο 2 της ημερήσιας. Έγκριση των πρακτικών 10-11 Απρίλη και 3-4 Μάη. Τα εγκρίνουμε και πάλι αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Δεν υπάρχει άλλη αντίρρηση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε τότε στις πληροφορίες. καταρχά για την στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα. Η συγγήτρια κυρία Μάισνερ. Αλλά πριν πάμε στην ψηφοφορία, να δούμε αν υπάρχει απαρτία. Να μετρήσουμε λοιπόν αν έχουμε απαρτία. Πάρτε την ηλεκτρονική σας κάρτα για την ψήφο. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της... Α, όχι, διακόπτει πρόεδρος, ναι, κυρία Δεκάμπ. Η κυρία Δεκάμπ, τι θέλετε, α, θέλετε να αλλάξετε θέση. Ναι, ναι, αλλάξετε θέση. Πολύ ωραία. Πέρας τις ψηφοφορίες, λοιπόν, όπως λέγαμε. Υπάρχει απαρτία. Οπότε, περνάμε στις ψηφοφορίες. Είσαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Γρήγορα. Παράγραφος 1. Ποιος είναι υπέρ. Συμβαστική. Διορθώνει το ρεπρό. Συμβιβαστική. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική τροπολογία 1 εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 6 απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 7 εγκρίνεται. Θέλετε όμως ηλεκτρονικό έλεγχο, έτσι, να ψήφισουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 15 κατά, δεν έχουμε αποχές, οπότε η τροπολογία του κυρίου Ρικέ εγκρίνεται. Τροπολογία 9, προχωράμε. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 60. Υπέρ της 60. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 60 εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 17 εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 3 εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές η 43 εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές η 4 εγκρίνεται συνεχίζουμε 24 υπέρ κατά αποχές η τροπολογία 24 απορρίπτεται η τροπολογία 25 28 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, η τροπολογία 28 απορρίπτεται. Τροπολογία 65 υπέρ, κατά, αποχές, η τροπολογία 65 απορρίπτεται. Θα ελέξουμε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. υπέρ 21 κατά 18. Κυρία Ρεβό, καλά κάνατε που ζητήσατε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, η 5 εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, η συμβαστική 6 εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, η 7 εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές η συμβαστική 8 εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές η 55 εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές η συμβαστική 9 εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 67 υπέρ κατά εγκρίνεται νομίζω αλλά θα ελέξω λέει η πρόεδρος άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 67 πέρας της ψηφοφορίας Ξαναλέει πρόεδρος πέρα της πληροφορίας. 67 εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ξανακάνουμε γιατί δεν σκόνεται το χέρι ψηλά λέει η πρόεδρος. Ξαναρχίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 42. Πέρα της ψηφοφορίας. Η 42 εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64. Το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο τη τροπολογία 64. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται βεβαίω, λέει πρόεδρο. Δεύτερο τμήμα τη τροπολογία μου, λέει πρόεδρο. Ποιο είναι υπέρ. Α, δεν το ίδιο, λέει ο πρόεδρο. Κατά. Αποχέ. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας μου δεν εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Και τελική ψήφος, έκθεση στο σύνολό τη για την κυρία Μάσνερ. ψηφίζουμε για το σύνολο της έκθεσης. Ψήφισατε όλοι, πέρα τη πληροφορία, υπέρ 40. Μια ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κυρία Μέσνερ. Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίνεται η έκθεσή σας. Συγχαρητήρια. Και εποφελούμε της ευκαιρίας επειδή έχουμε εδώ μια αντιπροσωπεία. Αντιπροσωπεία που υποδεχόμαστε, καλωσορίσατε, είστε από την Γερμανία, γυναίκες πολιτικοί, 10 νομίζω, βρισκόμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών όπου οι γυναίκες προηγούνται εδώ Καλωσορίσατε λοιπόν και ευχαριστούμε και την κυρία Μέσνερ που σας προσκάλεσε στην Επιτροπή μας. Συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο. Ανταλλαγή υπόψη με τον Γενικό Συγητή για τον Προπολογισμό 2018, τον κύριο Ζίκφριντ Μουρεσάν. Πού είστε κύριε Μουρεσάν. Δεν έχει έλθει ακόμη ο συγητής μας. notre rapporteur. Δεδομένου ότι ο εισηγητής, ο Γενικό εισηγητής μα για τον προπολισμό δεν έχει έρθει ακόμη και δεδομένου ότι είναι και αρχή τη εβδομάδα. έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πέντε λεπτών. Ευχαριστώ. Mes chers 5 Πέρασαν τα πέντε λεπτά. Ο προσκεκλημένος μας είναι εδώ κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίζω λοιπόν τον κύριο Μουρεσάν. Κύριε Μουρεσάν, είστε εισηγητής. Μιλάτε γαλλικά, εξαιρετικά. Ο εισηγητής μα είναι ο γενικός εισηγητής για τον Γενικό Προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Οικονομικό του 2018. Ευχαριστώ που ήρθατε για μια γενική ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις δημοσιονομικές προτεραιότητες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σώβει μια σοβαρή αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια οικονομική αναταραχή. Πρέπει λοιπόν να προβούμε στις βέλτιστες επιλογές όσον αφορά τις δημοσιονομικές μας προτεραιότητες, δεδομένου ότι οι πολίτες εξαρτώνται από αυτές ακριβώς τις επιλογές, δημοσιονομικές επιλογές. Η συνεργασία της Επιτροπής μας με την Επιτροπή Προπολογισμών ήταν καθέναν εξαιρετική. Πάντα οι συζητήσει μα ήταν σε κλίμα επικοδομητικό. Για μένα προσωπικό είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να είναι ενωμένο σε κοινό μέτωπο ως προς το θέμα αυτό εναντί ενός συμβουλίου που πολλές φορές είναι δύσκολο να πείσουμε. Κύριε Μουρεσάν, ελπίζω να προσφέρω σωστά το όνομά σας. Έχετε 10 λεπτά για να μας εκθέσετε τις γενικές γραμμές του προπολογισμού. Όσον αφορά δηλαδή τον προπολογισμό του 2018. Πείτε μας ποια είναι τα πρώτα σας συμπεράσματα, οι πρώτες σας εντυπώσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε τον προπολογισμό του 2018, για τον οποίο είμαι γενικό ηγητή στην Επιτροπή Προπολογισμών. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Τον Μάρτιο εγκρίναμε με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια την έκθεση όσον αφορά τον προπολογισμό του 2018. Αυτή είναι και η πρόταση η οποία περιέχει και τι πολιτικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2018. Κατόπιν αυτό, περιμέναμε την Κομισιόν να υποβάλει σχέδιο προπολισμού βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων, τι οποίε παρουσιάζει σήμερα η Κομισιόν. Ο Επιτροπός Έτιγκερ στην Επιτροπή Προπολισμών σήμερα παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού, έτσι, πέραν των πολιτικών προτεραιοτήτων που ήταν γνωστέ, Από σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, είδαμε τα πρώτα νούμερα. Εννοείται ότι δεν είχαμε χρόνο για εις βάθος αξιολόγηση αυτών των προτάσεων, αλλά μπορώ να σας δώσω κάποια τουλάχιστον νούμερα. Όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, πρότεινα από τις αρχές του 2017 να ιεραρχήσουμε ως ε, πρώτες προτεραιότητες δύο-τρεις τομείς. Πρώτον, ανάπτυξη και θέση εργασίας. Δύο, ασφάλεια όλων των μορφών ε, ασφάλεια για τους πολίτες της Ένωσης. Αλλά το πρώτο που υποσχόμαστε στους πολίτες, επαναλαμβάνω, είναι θέσεις εργασία και ασφάλεια. Για το πρώτο, στον τομέα αυτών πρέπει να επενδύσουμε, ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο αξιόπιστη, πιο ισχυρή. Πιο ανταγωνιστική, επαναλαμβάνω. Επενδύουμε λοιπόν σε υποδομές, στην καινοτομία, στην υποστήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Αυτή ήταν εξ αρχής η πρότασή μου. Στις κατευθυντηρίες γραμμές αναμένουμε η Κομισιόν να δουλέψει το ορίζοντας 2020 ε, για το κόσμο, για το Εράσμος και το καθεξής. Ε, δεν είναι, ξέρετε, το Εράσμος μόνο πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάνουμε τους νέους μας πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά. Έρευνε δείχνουν ότι 65% των εργοδοτών εκτιμούν την διεθνή εμπειρία αυτών των νέων ανθρώπων κάθε φορά που προσλαμβάνουν. Ζητήσαμε λοιπόν αυτά ακριβώ από την Κομισιόν. Τι έκανε η Κομισιόν στο πλαίσιο του σχεδίου προπολογισμού για το Horizon 2020 προτείνουν αύξηση 7% για το Connecting Europe, το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη 8% και για το Erasmus 9%. Για το COSME Έχουμε μικρή μείωση σε σύγκριση με το τρέχον έτος, είναι 9% η μείωση αυτή. Πέρσι όμως το έτος ήταν εξαίρεση γιατί είχαμε αυξήσει πάρα πολύ τον πολιτισμό. Για το κόσμο σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τους αριθμούς με μεγαλύτερη προσοχή για να δούμε αν πραγματικά όλα αυτά αρκούν για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το μηχανισμό σιδεών στην Ευρώπη ε, έχουμε μια αύξηση 8,7% σε δεσμεύσεις και 8,5 σε πιστώσεις πληρωμών. Στα μεγάλα πρόγραμματα υποδομών 0,1 συν η μεγαλύτερη αύξηση για το ίτερ 27%, 5,5 το Κοπέρνικους και 9,6 μείωση στο Έγνος και Γαλιλαίο, το πρόγραμμα των δορυφόρων. Εκεί οι πληρωμές αυξήθηκαν παρόλα αυτά 0,1%. Αυτά είναι τα νούμερα που έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον, Βάση, επαναλαμβάνω, τη εισήγη του κυρίου Έτιγκερ πριν από τρει ώρε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε έτσι μια πρώτη εικόνα. Θα μελετήσουμε τα νούμερα αυτά φυσικά περαιτέρω. Δεύτερη προτεραιότητα, ασφάλεια για του πολίτε εναντί ε, ατυχημάτων και απειλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει του ελέγχου στα σύνορα, την ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων στην Ευρώπη δεδομένου ότι έχουμε αρμοδιότητα για τη δικαιοσύνη και τις αριστικές υποθέσεις, θέλουμε να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ανθρώπων, θα αυξήσουμε λοιπόν τους σχετικούς προϋπολογισμούς και την στελέχωση της ε, Europol, Frontex, EASO και της Ιουλίσα και επίσης στην έρευνα για την άμυνα έχουμε 40, εκατομμύρια επιπλέον για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε καλύτερα τις συνέργειες μεταξύ άμυνας και έρευνας. Να σταματήσουμε λοιπόν να δαπανούμε για προγράμματα έρευνα στην άμυνα ανεξάρτητα από όλα τα άλλα. Έτσι, ξοδεύουμε μία φορά και καλύπτουμε όλου του τομεί και φυσικά τα αποτελέσματα, τα πορίσματα είναι κοινά μεταξύ όλων των εταίρων. Για να εξασφαλίσουμε περισσότερη ασφάλεια στα σύνορα, πρέπει επίση να διασφαλίσουμε ότι στην άμεση γειτονία μα, που στην Ανατολή ειδικά, οι γειτονέ μα, οι γειτονικέ χώρε που έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία και που βαδίζουν στον δρόμο τη Ευρώπη και που ήρθαν πίεση του Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτές οι χώρε λοιπόν χρειάζονται υποστήριξη. Είναι οι χώρε οι αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της εισόδου μεταναστών, της μαζικής εισόδου μεταναστών. Βάσει μελέτης είναι πιο ασφαλές και πιο οικονομικό και πολιτικά πιο εύπεπτο να γίνει η διαχείριση των ε, μεταναστών και των προσφύγων στην Ιορδανία, το Λίβανο, ε, παρά όταν φτάσουν πια στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει αυτών, να επιστήσω την προσοχή σας, την αναθεώρηση του επτάετους πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου, έτοιμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμβαστική πρόταση. Εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε αρκετή δουλειά. Άλλωστε, οι συνάδελφοι που είναι και στην Επιτροπή Προπολογισμών γνωρίζουν ότι εγκρίναμε την συμφωνία αυτή με μεγάλη ταχύτητα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Α κάνει τώρα ό,τι πρέπει να κάνει και το Συμβούλιο. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο προ το παρόν έχει φρενάρει την έγκριση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κοιτάξτε, μέχρι τις 8 Ιουνίου, αν συνεχιστεί αυτή η ε, παρουσίαση προσκομμάτων, το, το καταλαβαίνουμε με τις Βρετανικές εκλογές, αλλά από εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά θα είναι ε, αλλιώς πολύ δύσκολο να καταρτήσουμε γέρος προπολογισμό για το 18, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 18. γιατί ακόμα πατάμε πάνω στις αποφάσεις του 13. Πάντως ήδη η Κομισιόν πιέζει το Συμβούλιο, έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη σχετική έγκριση. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη από το Ηνωμένο ότι έχουν την πρόθεση να μην εγκρίνουν την αναθεώρηση αυτή του πολιτού, του δέλτα, Άρα θεωρώ ότι αμέσως μετά τις Βρετανικές εκλογές και το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει την θετική του ψήφο. Πάντως συνεχίζουμε να πιέζουμε το Συμβούλιο έτσι ώστε το Συμβούλιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τώρα, όσον αφορά τα δικά σας θέματα, πέρα από το Connecting Europe, το μηχανισμό Σύνδεων στην Ευρώπη, είπα ότι για μας αποτελεί προτεραιότητα, το είχατε πει και εσείς, ανταποκρίθηκε η Επιτροπή, προτείναμε αύξηση των σχετικών κονδυλίων, Πέραν αυτών, λοιπόν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διαδικασιών οι οργανισμοί της ΕΕ δεν θα πληγούν από περαιτέρω μειώσεις. Δεν θα μειωθεί το προσωπικό αυτών των οργανισμών το 18. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό έχουμε ενσωματώσει και εμείς τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονήσαμε τον Μάρτιο. Αυτό σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι φτάνω στο τέλος της εισηγησής μου. Είμαι εδώ βεβαίως για να συζητήσουμε με τους βουλευτές. Έχετε ήδη ένα σχέδιο προπολισμού. Έχετε μεγάλη πείρα σε τέτοια θέματα. Εγώ εδώ, αν θέλετε, να συζητήσουμε όπως μπορώ να συζητήσουμε και με τους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολισμού. Ευχαριστώ πάντως για την πρόσκλησή σας και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μουρεσάν, δίνω τον λόγο στον συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Τοσενόφσκι, που θα μας δώσει την οπτική γωνία της Επιτροπής μας. Παρακαλώ και μετά θα δώσω το λόγο στους ε, σκιώδες, αλλά έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το λόγο. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Μουρισάν για την παρουσίαση που μας έκανε και για την έγκαιρη ενημέρωση που μας έδωσε σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση του προπολογισμού. Ως ε, εισηγητής ε, για λογαριασμό της Επιτροπής Μεταφορών θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για μας και τα οποία ε, περιλαμβάνονται και σε όλες τις προτάσεις που κάνει η Επιτροπή μας. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το εργαλείο του Connecting Europe. Επιχαίρουμε το γεγονός ότι θα έχει πλέον ε, περισσότερα κονδύλια καθώς ε, πράγματι αυτή η διευκόλυνση αποτελεί ένα από τα εργαλεία χρηματοδότησης των έργων στις μεταφορές. Στο παρελθόν είχαμε διαπιστώσει τόσο μετακινήσεις αν θέλετε κάποιων κοντιλίων, αλλά και κάποιες επερικοπές, οπότε ε, με χαρά μας ε, διαπιστώνουμε ότι επαναρχόμαστε τώρα σε ένα αξιοπρεπές εντός εισαγωγικών επίπεδο κοντιλίων ε, για την πρικοδότηση του Connecting Europe Facility. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να καταστήσουμε τον τομέα των μεταφορών πιο ελκυστικό για του ιδιώτε χρηματοδότε, την ιδιωτική χρηματοδότηση. Υπάρχουν και ενισχύσει οι οποίε χορηγούνται και οι οποίε μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο τρόπο για την ε, παροχή επενδυτικών ευκαιριών στι υποδομέ. Μία από τι προτεραιότητέ μα είναι ενίσχυση των σιδηροδρομικών ε, του σιδηροδρομικού δικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό σχετίζεται με αυτά που αναφέρατε εσείς, δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο προωθούμε και την, ε, τις ε, θέσεις εργασίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και τις ε, σταθερές θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν οι σιδηρόδρομοι ω τέτοιοι σημαίνουν περισσότερη Ευρώπη και σημαίνουν ισχυρότερη υποδομή. Είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα έγνος και Γαλιλαίο, δηλαδή τα δύο μας ε, δαρυφορικά συστήματα, καλύτερα στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε αυτά τα δορυφορικά προγράμματα και νομίζω πως μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλή βάση για αξιοποίηση στα συστήματα πλοήγησης στις μεταφορές και μάλιστα ε, για συστήματα πολύ ακριβούς πλοήγησης. Αποτελούν ταυτόχρονα πολύ καλές ε, επιχειρηματικές ευκαιρίες και Ε, οι εν λόγω δορυφόροι δίνουν και σήματα χρόνου, time signals. Όμως δεν κατάλαβα σωστά τα όσα είπατε σε ό,τι αφορά τον Καλιλαίο και την ε, μείωση εκεί των κοντιλίων. Εάν σας κατάλαβα σωστά. Τα δορυφορικά συστήματα ενισχύουν την ε, πολυτροπικότητα των μεταφορών κατανέμοντας ε, πιο ισορροπημένα τις ε, ροές των μεταφορών και έχουν και μια σειρά από περαιτέρω ωφέλη. Εγώ είχα την ευκαιρία να διαβάσω τις ε, προτάσεις των πιλωτικών προγραμμάτων που είχαν Ε, προήλθε από τη δική μας επιτροπή, δηλαδή 23 ε, διαφορετικά project ε, με συνολικό προπολογισμό της τάξης των 28 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε πως αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εφαλτήριο τόσο για την ενίσχυση υφιστάμενων προγραμμάτων όσο και για την έναρξη καινούριων. Αναμένω με ενδιαφέρον τις περαιτέρω συζητήσεις που θα έχουμε και με εσάς και με του σκιώδει εισηγητέ ε, και βέβαια θέλουμε να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα δυνατά κονδύλια για τον επόμενο προπολογισμό. Ευχαριστώ, κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Μουρισάν, σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Είναι θετικό το γεγονό ότι ο κύριο Σόντιγκερ ενέκρινε σήμερα το πρωί με βάση τα όσα άκουσα την πρόταση προπολογισμού από την πλευρά λοιπόν των ε, μεταφορών, ε, το πιο σημαντικό είναι, νομίζω, ότι θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο η, τα όσα προβλέπονται διατάξεις δηλαδή της ενδιάμεσης ανθεώρησης περιλαμβάνονται σε αυτό το προπολογισμό όπως είχε υποσχεθεί ο κ. Σότινγκ Είχε ανακοινώσει δηλαδή στο παρελθόν ότι θα περιλάμβανε αυτές τις διατάξεις ε, και πρέπει να το διαφανίζουμε. όχι μόνο για το Connecting Europe Facility, για το ΣΕΦ, αλλά και επειδή είχαμε ε, κάποια μεταφορά κονδυλίων από τα επενδυτικά προγράμματα στο, ε, Και ο συνάδελφος εδώ αναφέρθηκε και στα δορυφορικά μας ε, συστήματα, ε, όπως το έγνωστο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως γνωρίζετε δεν έχουμε πλήρη κάλυψη δηλαδή όλης της Ευρώπης από αυτά τα δορυφορικά συστήματα και γι' αυτό χρειαζόμαστε και περαιτέρω χρηματοδότηση ώστε να καλύψουμε τη Βόρεια Αφρική, δηλαδή τη Νότια και Νοτιονοτή Ευρώπη και τη Βόρεια Ουκρανία. Δηλαδή εδώ ε, δεν αναφέρομαστε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στην πολιτική γειτονία σε ό,τι αφορά δηλαδή, την κάλυψη, την δορυφορική από αυτά τα συστήματα. Οπότε, εάν αυτή η πτυχή δεν περιλαμβάνεται στον προπολογισμό, εμεί θα προτείνουμε κάποιε ε, ε τροπολογίε, ώστε να ασφαλίσουμε αυτά τα συμπληρωματικά κονδύλια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δαπανηρό, γύρω στα 10 εκατομμύρια, σχεδόν τίποτα δηλαδή. Και αυτό ξαναλέω για να καλύψουμε την ε, Ανατολική Ευρώπη αλλά και το ανατολικό εκεί το πέμα. Και αναμένω ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε τις συνδρομικές μεταφορέ και ειδικότερα το Interrail. Ήδη έχει ανακοινωθεί παντού έτσι ότι το υποστηρίζετε. Οπότε είναι σημαντικό να το κάνουμε στην πράξη. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε. Θέλετε να ασχολείστε εσεί Ναι, ίσω να απαντήσω. Τώρα, γιατί είχαμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. η ενδιαμέση αναθεώρηση του πολιτού του μισονομικού πλαισίου. Αυτά περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προπολογισμού. Είδαμε το πρωί τα ποσά για το Connecting Europe Facility, για το Erasmus, για το 2020. Τα είδαμε αυτά. Και θέλουμε ακριβώς να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα κονδύλια μέχρι την διάμεση αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου. για την ανατολική μας γειτονιά και την Ουκρανία. Το μόνο που ξέρουμε είχαμε μια αύξηση 8,9% για την ανατολική μας γειτονία, δηλαδή 46 εκατομμύρια ευρώ σε απόλυτους όρους. Δεν ξέρουμε λεπτομερώς πώς θα διαρθωθούν αυτά τα χρήματα, αλλά θα αφορά και την Αφρική αλλά και την Ουκρανία και τα προγράμματα και θα το παρακολουθούμε. Για τον Είναι 9,6 μείωση στο σχέδιο της Κομισιόν, αλλά πρέπει να το δούμε μαζί και να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτό όντω είναι ενσχετικό για σας. Και αν αυτό δεν είναι αποδεκτό από την Επιτροπή σας, να το ξέρουμε και να το μεταφέρουμε στην Κομισιόν. Το ίδιο για τον Ιντεραήλ. Δεν είναι μυστικό ότι ο πρόεδρος της ομάδας μας πέρσι είπε στην απάντηση στην κατάσταση της Ένωσης ότι ο κάθε πολίτης της Ένωσης άνω το 18 θα πρέπει να έχει ένα ελεύθερο στήριο Interrail από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εγώ είπα θα το σπίσω αυτό, θα το εντάξω στις κατευθύνσεις γραμμές και στις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. για τον προϋπολογισμό του 18, ώστε να βρούμε τους πόρους για το 18 κιόλας και πράγματι αυτό το ανακοινώσαμε δημοσίω. Τώρα, ο Πίτροπος Έντικερ λέει το εξή ότι είναι έτοιμος αρχικά να χρηματοδοτήσει το Interrail. Δεν θέλει όμως αυτό να θέσει σε κίνδυνο να εξελίξει και υπάρχοντα προγράμματα. Γι' αυτό ακριβώς κατευθυντήρηση είπαμε ότι θέλουμε να το χρηματοδοτήσουμε βάσει ενός μακρόπνου σχεδίου σταθερού και προβλέψιμου. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ξεχωριστή γραμμή του προπλογισμού ξεχωριστή δηλαδή από το Εράσμους, ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο το Εράσμους και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα νομοθετική βάση, κάτι το οποίο από την Επιτροπή και ο να Επίτροπος Ναυράτσης για την νεότητα ή από την Επιτροπή και τον Αρμόδιο Επίτροπο για τις πρέπει να προταθεί. Αν πάντω οι συνάδελφοι εδώ, η πλειοψηφία συναδέλφων εδώ στην Επιτροπή Τραν το μεταφορών υπέρ αυτού του Interrail και τη πρωτοβουλία, τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει μια πρόταση για την κατάλληλη νομική βάση γι' αυτό. Τι τελευταίε μέρε πάντω ήρθα σε επαφή με την Κομισιόν και η ότι ακόμα δεν έχουν καταθέσει πρόταση για το Interrail στο τωρινό σχέδιο προπολογισμού, επειδή δεν έχουν την απαραίτητη νομική βάση. Υπάρχει ένα μικρό πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε φέτο υποβλήθηκε πέρσι και ξεκίνησε φέτο, αλλά δεν είχαμε αυτό κατά νου. Η Κομισιόν λοιπόν λέει ότι δεν είχα νομοθετική βάση και αυτό δεν έκανα συγκεκριμένη πρόταση, αλλά σπάμε στους επιτρόπους και στην Επιτροπή μετά από τη συνάντησή μας εδώ, να δούμε αν έχει προχωρήσει το θέμα την νομική βάση και να δούμε αν αυτό μπορούμε να το εντάξουμε στις διαπραγματεύσεις και στον τριμερή διάλογο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο ώστε να εγκριθεί για τον επόμενο προπολογισμό του χρόνου δηλαδή. Μπορούσε να βράτσει οι δύο επιτροποί είναι αρμόδιοι, να δούμε κατά πόσο λοιπόν αν υπάρχουν εξελίξεις για την νομική βάση. Πρέπει όμω τώρα ειλικρινά να δούμε και το πόσο μεγάλα είναι τα διαθέσιμα ποσά. Η Κομισιόν είπε ότι το περιθώριο αφορά 51 εκατομμύρια ευρώ από τον τωρινό προπολογισμό. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά. Όμως εμείς θα θέλαμε κάτι πέραν του τωρινού πιλωτικού προγράμματος που έχουμε για φέτο, όπως λέγαμε, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το Interrail, το ελεύθερο, το δωρεάν ειστήριο δηλαδή, για όλου του άνω των 18. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν για να εξετάσουμε τις νομικές βάσεις, ώστε να έχουμε προβλέψιμη και σταθερή χρηματοδότηση για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Συνεχίζουμε. Με τους υπόλοιπους ομιλητές, ο κ. Σαρτούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μουρεζάν, καλώς Έχω την χαρά να σας αναφέρω την ε, δήλωση της Σκιώδου του κ. Γκραπίνη. Ευχαριστώ καταρχάς όλους τους εμπλεκόμενους για την καλή συνεργασία και όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν πλοκές προτάσεις και προπαρασκευαστικές δράσεις. Για τις 28 παρασκευαστικές δράσεις και τα πλοκές προγράμματα για τον τουρισμό και τις μεταφορές, και μεταξύ αυτού έχουμε 17 νέα. Έχουμε πέντε αφορούν τον τουρισμό, μεταφορές γενικότερα. Κάποια από αυτά συνεχίζουν προϋπάρχοντα προγράμματα στον τομέα ιδιαίτερα των μεταφορών. Προτείνουν λοιπόν 7 πιλωτικά προγράμματα και το συγκεκριμένο που προτείνει η κυρία Γκραπίνη αφορά την πρόθεση του τοπικού τουρισμού στην Ευρώπη. συνυπογράφουν και η Γκουε και η ΑΛΤΕ αυτή την πρόταση μας πολιτικές ομάδες, ώστε να προωθηθούν πρωτοβουλίες τοπικής φύσης για τον τουρισμό, δηλαδή τοπικά Airbnb σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και συνεργασία σε διάφορα σημεία όσον αφορά τις μεταφορές μέσα εκπόνησης διαφόρων προγραμμάτων που θα περιέχουν και ένα διαδραστικό οδηγό. Υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι εδώ. Έχουμε και πέντε νέες παρασκευαστικές δράσεις στο PA1, τρεις στο τουρισμό και δύο στις μεταφορές. Προτάθηκε να συνεχίσουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις που ξεκίνησαν πέρσι στον τομέα θαλάσσιων ε, μεταφορών, κάτι που αφορά την εκπαίδευση των πληρωμάτων. Μετά έχουμε επίσης και κάτι που πρότειναν το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι και τρεις πρωτοβουλίες ή προτάσεις των σοσιαλιστών. Ο αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών πρότεινε ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό και τις ευφυείς μεταφορές και συστήματα ευφυών μεταφορών και ποδηλασία. Ο τουρισμός στις μεταφορές είναι ένα νέο στοιχείο τουρισμού επηρεάζει και την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη και είναι σημαντικό να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια σε αυτό το πεδίο επειδή θα μπορέσει να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της ύφεσης και της ανεργίας. Η ποιότητα και η διαφοροποίηση των υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιώνονται συνεχώ ώστε να διατηρήσουμε την ηγετική θέση της Ευρώπης ως τουριστικό προορισμό. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή και τους σκιώδες για την καλή συνεργασία και όλους τους αδέλφους που υπέβαλαν πιλωτικές προτάσεις, πιλωτικά προγράμματα και προπασκευαστικές δράσεις. Και ελπίζω να καλά, όλα να πάνε καλά στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ρωτού. Ο κύριος Λίνσκα, έχετε το λόγο. Ε, χαιρόμαστε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, ε, κύριε Μουρεσάν. Ε, καταρχήν, ε, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που αναφέρατε, δεν νομίζω πως μπορεί να διαφωνήσει ε, κανείς μαζί σας και θα πρέπει να σας υποστηρίξουμε. Αν δούμε δηλαδή ε, τα όσα μας απασχολούν στην Επιτροπή Τραν ε, των Μεταφορών, ε, πράγματι οι δύο προτεραιότητες που έχετε ονομάσει είναι συνδεόμενες. Δηλαδή από τη μία πλευρά οι μεταφορές αποτελούν κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά από την άλλη πλευρά η ασφάλεια ε, και από ατυχήματα και από εξαιρετικέ επιθέσει αποτελεί αναπέρασπαστο μέρο αυτή τη ε, πολιτική. Οπότε θα πρέπει ε, να δούμε πώ θα κατανεμηθούν τα κατάλληλα κονδύλια για αυτέ τι δύο πτυχέ τη ασφάλεια προκειμένου να αξιοποιηθούν με τρόπο ο οποίο θα αποβεί προ όφελο των μεταφορών. Ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και είναι σημαντικό όχι μόνο λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα εδώ στην Ευρώπη, αλλά και επειδή αποτελεί ένα ε, μεγάλο πρόβλημα για όλους μας ε, και τους αερολιμένες μας ως προς το πώς θα το αντιμετωπίσουν και επειδή δεν θέλουμε να περιπλέξουμε και τις ζωές των πολιτών μας είναι ακριβώς η ε, προτεραιότητα που αναφέρεται οπότε νομίζω πως ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή να συνδυάσουμε τις δύο προτεραιότητες καλύτερα μαζί τους. Τώρα σε ό,τι αφορά την ανακοινωθήσα αύξηση των κονδυλίων ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Connecting Europe ε, Facility, δηλαδή το σημείο 7. Σίγουρα είναι θετική αυτή η αύξηση, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, ε, ποια ήταν και η αύξηση που έγινε κατά τελευταία περίοδο. Ενδεχομένω δηλαδή να πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσει. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αποτελεί μια θετική εξέλιξη αυτή η αύξηση. Το ερώτημα που τίθεται για μένα είναι ε, ενδεχομένως μια σύγκριση του Interrail το οποίο ξεκίνησε ως ένα mega project, ως ένα έτσι έργο μεγάλων διαστάσεων, τεραστίων διαστάσεων, το οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι είχε προβλεφθεί ότι θα απέβαινε προς όφελος της εκπαίδευσης των, ε, των ε, νέων ή θα συνέβαλε για, στη δημιουργία του ενίου χώρου μεταφορών. Ε, και κατά κάποιο τρόπο εισάγει διακρίσεις γιατί υποστηρίζει μόνο ένα τρόπο μεταφορών, ένα μέσο μεταφορών. Οπότε υπάρχουν και αυτέ οι πτυχέ τι οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Δηλαδή, ε, ε, θέλουμε να επενδύσουμε κονδύλια σε ένα εργαλείο το οποίο έχει μια ισχυρή πολιτική διάσταση πράγματι, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα και να, τηρεί, να πληρεί και κάποια κριτήρια τα οποία ανέφερα μόλις τώρα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αποβαίνει ε, ε εις ε, άλλων χρήσιμων και επιτυχημένων project. Δεν θα ήθελα δηλαδή αυτή η αύξηση των κονδυλίων για το ίντερνετ να αποβεί σε μείωση των αντίστοιχων κονδυλίων για τα δορυφορικά ε, προγράμματα έγνωση και Καλλιλέο. Γιατί τα Έγνωση και Καλλιλέο αποτελούν επένδυση στο μέλλον. Και έχουμε και το ζήτημα πέραν των, ε, μεταφορών, δηλαδή των υπηρεσιών, αλλά και τη ασφάλεια αποτυχήματα και ασφάλεια από εξωτερικέ Οπότε νομίζω πως αντιλαμβάνεσαι το μήνυμα που θέλω να περάσω και εγώ και η ομάδα μας ή η Επιτροπή μας γενικά. Σίγουρα δηλαδή αν πληρεί το Interrail τα κριτήρια που ανέφερα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ε, αναφέρθηκαν και από κάποιου άλλου συναδέλφου ε, κάποια ζητήματα πέραν ε, ενό. Δηλαδή, ο συνάδελφο ε, του Ενώστη αναφέρθηκε στο ζήτημα των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά ενδεχομένω εκείνο που θα πρέπει να μα απασχολήσει και είναι η, ο συνδυασμό μεταξύ των διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων. νομίζω πω αυτό ο συνδυασμό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρία Κίλωνεν, παρακαλώ, λέει πρόεδρος. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κονέτσκα σκιώδους εισηγητρίας. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Πάντως θα ήθελα περισσότερη χρηματοδότηση για τις πολυτροπικές μεταφορές και θα ήθελα περισσότερη χρηματοδότηση για το μέλλον των σιδηροδρόμων που φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρούσα φάση. Στο πλαίσιο του, της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα της χρηματοδότησης της καινοτομίας και δι, η δημίωση των εκπομπών ανθρακά. Εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, αξιοπρεπή χρηματοδότηση όπω και η χρηματοδότηση για, τον περιορισμό των εκπομπών γενικότερα, την αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος κλπ. Αυτά αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, αλλά και ανθρώπινους πόρους. Φυσικά πρέπει να παρακολουθούμε τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών. Αυτά προς το παρόν από μένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ξαναβλέπω τον ε, εισηγητή. Τα είχαμε ξαναπεί. Λοιπόν, προτεραιότητες. Ασφάλεια και θέσει εργασία. Ναι, γιατί όχι, συμφωνώ. Αλλά όταν λέμε θέσει εργασία, τι ακριβώ εννοούμε. Θέλουμε θέσει με διάρκεια. Θέσεις για το μέλλον. Γι' αυτό έλειπε εν μέτρο τιμή. Όταν ε, συζητούσαμε και είχατε προτείνει τι γνωστέ προτεραιότητε. και αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Ποιο είναι το μέλλον των θέσεων εργασία για εμά τους Ευρωπαίους. Στον προπολογισμό μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα και επειδή είμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών. Ναι, τι είδου υποδομές θα δημιουργήσουμε, τι θα προαγάγουμε. Όταν λέμε υποδομές, ε, εννοούμε κατασκευέ που θα είναι εδώ μαζί μας για πολλές δεκαετίες. Και αυτό που είπε η κυρία Κιλονέν. Δηλαδή, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους όσον αφορά το κλίμα, να φροντίσουμε και οι υποδομές να συνάδουν με τον στόχο αυτό. Δηλαδή, η Ευρώπη στο G7 καλά τα λέει σχετικά με το Παρίσι και την εφαρμογή του, όμως να φροντίσουμε ότι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνουμε όλα σωστά. Δηλαδή, προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργία θέσεων εργασία να κρατηρούν προς τον ίδιο στόχο. Αυτό είναι το βασικό μέλημα. Θα ήθελα λοιπόν να έχετε πει λίγο περισσότερες στην εισαγωγή σας για το θέμα, αλλά νομίζω ότι μαζί θα πετύχουμε το ζητούμενο. Γι' αυτό και προτείνουμε κάποιες γραμμές στον προπολογισμό και κάποια πιλωτικά προγράμματα, στην εκπαίδευση, ε, να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει, τι σημαίνουν αεφορικές μεταφορές, ας πούμε, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, από την ε, εκπαίδευση, για, αν θέλουμε να έχουμε έναν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Αυτό είναι και ο στόχος του προπολογισμού, ο ρόλο, αν θέλετε, του προπολογισμού. Αυτά θα ήθελα λοιπόν να προσθεθούν στον προπολογισμό. με βέβαιο ότι θα τα πετύχουμε σε συνεργασία με εσά ω εισηγητή. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε μια παρατήρηση. Άκουσα τον εισηγητή και τις προτεραιότητες, απασχόληση, ασφάλεια, ναι. Ευλογή και επενδυτή στόχη. Άκουσα και το έρασμος, το έρασμος για την απασχόληση. Όντως, πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Που πραγματικά, πέρα από τη σχετική γραφειοκρατία, είναι πρόγραμμα με προπολισμό και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια. Ε, αυτό πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγράμματα με τα οποία οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν την προσθεμένη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θεωρώ πάντως ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με την εξή έννοια. Ήμουν Πρίτανης ε, σχολή ε, Γλωσσών όπου διδάσκαμε 27 ξένες γλώσσες και πολιτισμούς και διαπιστώναμε ότι είναι πολύ χρήσιμο φυσικά για τους Γάλλους που μαθαίνουν Ισπανικά να μπορούν να πάνε έξι μήνες να, στη Μαδρίτη ίσως και περισσότερο ε, εάν η οικονομική κατάσταση των γονέων τους το επέτρεπε και αντιστρόφως οι Ισπανοί φοιτητέ έρχονται στην Γαλλία κλπ. Για να έρχονται σε επαφή με την ίδια τη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται αυστηρότητα ως προς τα κριτήρια διότι και στο Έρασμος αλλά και σε άλλα προγράμματα στα οποία εμπλέκεται η τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση ε, η τάση ήταν ο ούτως επίν πανεπιστημιακός τουρισμός. Δηλαδή, καλό είναι να ναι, καλό είναι να ζεις στο εξωτερικό, αλλά το θέμα είναι να παρέχεται εκπαίδευση και ειδικά επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μάλιστα επίπεδου. Όποιος πηγαίνει λοιπόν στο εξωτερικό να έχει τις απαραίτητες ελάχιστες γνώσεις και την ελάχιστη ικανότητα χρήσης της γλώσσας της χώρας στην οποία πηγαίνει ή όπου εν πάση περιπτώσει ε, θα παρασχεθεί σχετική εκπαίδευση. Οπότε δεν λέω καλός και ο τουρισμός αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Είμαι υπέρ λοιπόν του προγράμματος, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν βλέπω σε ό,τι με αφορά κάποια άμεση θετική επίπτωση στην αγορά εργασία, γιατί η ενεργία έχει άλλα αίτια, πολύ σημαντικά, άλλη φύση. Α πούμε, η κατάργηση των δασμολογικών εμποδίων έχει ω αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι μα να ανταγωνίζονται ευθέω εργαζομένους που παιρνουν μισθου μισθούς 20-30 φορέ ε, μικρότερους. Αυτό είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε τώρα μέσω του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά πάντως την εκπαίδευση, ναι, είμαι υπέρ των ανταλλαγών με το εξωτερικό, με την προϋπόθεση όμως επαναλαμβάνω ότι τα κριτήρια θα είναι συγκεκριμένα και αυστηρά και το πρόγραμμα και ότι μάλλον στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση ε, οι νέοι με τα απαραίτητα προσόντα και τις ελάχιστες απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκόλνης, εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ για τη γνώμη σας όσον αφορά το πρόγραμμα Έρασμος, αλλά ε, δεν το χειρίζομαι εγώ, έτσι, το πρόγραμμα Γκόλνης. Νόμιζα ότι θα μιλούσατε για το Interrail. Γκόλνης. Όχι, το Erasmus δεν το έθεσα. Εγώ ο εισηγητής το έθεσε προηγουμένως. Και αναγκαστικά ακολούθησα και εγώ. Το Erasmus αφορά και τις μεταφορές και τον τουρισμό. Μιλάμε για διεθνείς ανταλλαγές, έτσι δεν είναι. Και δι των νέων. Εξού και η παρέμβασή μου. Πρόεδρος. Ακουστήκατε, κύριε Γκόλνης, κύριε Στεκά. Πρόεδρε, καλώς ορίζω τον Ζίγκφριτ στην Ομίγυρη. Τρία πράγματα. Πρώτον, για το για τα ευρωπαϊκά μάλλον ταμεία στρατηγικών επενδύσεων ε, και το ένα και το δύο ποια είναι η χρησιμότητά τους ε, έχουμε δάνεια προκειμένου και έχουμε και επιχορηγήσεις διευκολύνουμε έτσι τις επενδύσεις και με ποιο τρόπο συγκεκριμένα και πόσο διευκολύνουμε τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Υπάρχουν πολλές πρακτικές δυνατότητες, δεν υπάρχει καμία εμφόλια. Α πούμε και, και το Ταμείο Συνοχής, στο, στον τομέα των μεταφορών συγκεκριμένα. Ε, πώς το βλέπει αυτό η Επιτροπή Προπολογισμών, μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Και κάτι άλλο, εκ του προχείρου, να μου επιτρέπετε, σχετικά με το Interrail. Δεν είμαι υπέρ των εμποδίων και των φραγμών εδώ, αλλά αν μας λέτε ότι δεν υπάρχει γραμμή στον προϋπολογισμό, αυτό σημαίνει ότι δεν το θέλουμε τελικά. Δεν το θέλετε. Ε, τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν τραγικά πράγματα στον πλανήτη και προσθέσαμε γραμμές στον προπολισμό για να κάνουμε κάτι. Δεν θέλω να αρθώσω προς κόμματα, αλλά λέω προς τον κύριο Λίτσκε, προς τον κύριο Λάμπστορφ, ότι η αίσθηση που έχουν ότι κάτι λάθος έχει γίνει εδώ. Το λέω και προς την κυρία Χάρμς αυτό. Γιατί θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν και δεν ξέρω πραγματικά τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ κύριε Φαντεκάμπ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κράμερ. Σας ευχαριστώ και εγώ την, ε, για την παρουσίαση. Το γεγονό ότι είμαστε υπέρ τη δημιουργία θέσεων ε, και υπέρ τη ανάπτυξης είναι ένα τροπάριο, αν θέλετε, που το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, αλλά το ακούμε εδώ και χρόνια, χωρίς να γίνονται πολλά. Αλλά υπάρχουν κάποια παραδείγματα που είχαμε θετικά αποτελέσματα. Ε, για παράδειγμα, είχαμε ε, ένα συγκεκριμένο τρέμα στη Γερμανία, ε, το οποίο έπρεπε να κλείσει το 1992 αλλά ε, τελικά δεν έκλεισε ε, και σήμερα έχει χιλιάδες παραπάνω επιβάτες και μάλιστα έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Και από 4.000 τώρα ε, επιβάτες ένα άλλο, επιβά... ένα άλλο δρομολόγιο έχει πάει σε 23.000 επιβάτες ε, σήμερα οπότε ε, πραγματικά βλέπω να επενδύουμε για κάποια, σε κάποια μεγάλα project και τελικά δεν τους δίνουμε την κατάλληλη σημασία. Για παράδειγμα υπήρχε το Λεόν του Ρίν 12 δισεκατομμυρίων ευρώ και τελικά το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι θα είναι 26 και ότι από, ε, απλά η αύξηση των τρένων από 3 τεζεβέ θα ήταν 5. Και τι κάνουμε τώρα. Ε, στέλνουμε απλά δηλαδή έναν, ε, ένα τρυπάνι, θέλετε, ένα είδο μετροπόδικα, το οποίο απλά σκάβει μέσα στο βουνό για κάποια χρόνια. Πόσε θέσει εργασία δηλαδή δημιουργεί κάτι τέτοιο. Ε, πραγματικά ποτέ όταν σχεδιάζουμε τέτοιο είδου project δεν το λαμβάνουμε υπόψη τελικά, δηλαδή πιο αντίκτυπο έχουν και σε επίπεδο θέσεων εργασία. Προφανώς είμαστε περήφανοι για κάποια project ε, τα οποία λαμβάνουν χώρα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και πόσε θέσει εργασία δημιουργούν. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω, ε, ε ποια προτεραιότητα δίνεται σε μικρότερα project, τα οποία για παράδειγμα πραγματικά αυξάνουν κατά 95% για παράδειγμα τον αριθμό των επιβατών σχέση με το, ε, με το παρελθόν. Για παράδειγμα, στη Γερμανία ε, τα τρένα τα νυχτερινά ε, έχουν καταργηθεί ουσιαστικά. Ε, ε, επειδή θεωρήθηκαν ακριβώς ότι δεν, είναι, δεν ήταν αποδοτικά πλέον. Αντιθέτως όμως στον ε, τομέα των αεροπορικών έχουμε μια σειρά αποπτήσεις οι οποίες βρίσκονται ακριβώς στην διακατάσταση Ουσιαστικά δηλαδή όμως εκεί δεν συμβαίνει κάτι ενώ στα τρένα ακριβώς θεωρήθηκε ότι ε, παρότι είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικά δεν έγινε τίποτα. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Η κυρία μας. Μάλιστα, συγγνώμη. Ναι, ε, πολλά ήδη αναφέρθηκαν ε, ήδη εδώ, δηλαδή ότι ε, πράγματι, το, για παράδειγμα, το ΣΕΦ θα πρέπει να ενταχθεί και ανήκει στο ΤΕΝ. δηλαδή, πράγματι είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτά τα δίκτυα προ όφελο τη ολοκλήρωση τη Ευρώπη και βέβαια δεν θα πρέπει να γίνουν περικαπέ σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για τα δορυφορικά προγράμματα. Πάντω, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το ίντερ, γιατί αναφέρθηκε από, και από συναδέλφου και από τον Αλεξάνδρα Λάμπστοφ, τον αγαπητό μου φίλο. Αυτός, ε, ε, αυτή η ιδέα που ε, Αναφέρθηκε ότι δηλαδή θα δίνουμε στους 18χρονους ε, δωρεάν ε, ένα ε, τέτοιο εισιτήριο Interrail. Είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαστε αγιοβασίλειδες εδώ, δηλαδή αυτό θα κοστίσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα συμφωνήσω εδώ με τον συνάδελφο. Έχει τελικά προστιθέμενη αξία. Ποιο θα μπορέσει να αξιοποιήσει κάτι τέτοιο. Τι θα συμβεί με του ανθρώπου που ζουν σε νησιωτικέ περιοχέ, τι θα συμβεί με του ανθρώπου που δεν έχουν τη δυνατότητα να διανεκτερεύσουν κάπου αλλού, αν αξιοποιήσουν το Interrail. Οπότε πραγματικά είναι σημαντικό να δούμε από την Επιτροπή σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιτύχουμε κάτι για να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στου ε, νέου μα, αλλά σε καμία περίπτωση έτσι απλά να δώσουμε ένα δώρο Interrail δεν νομίζω πω είναι η σωστή άγουσα. Ευχαριστώ. Κύριε Ισηγητά, εσείς διαδραματίζετε εδώ σήμερα έναν ρόλο κλειδί και είστε στραμμένος στο μέλλον και στις προοπτικές και το λέω αυτό με την, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε δεμένοι στο βραχυπρόθεσμο. Δύο πράγματα λοιπόν θέλω να πω. Πρώτον, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ο προϋπολογισμός είναι πλέον ένας σχετικά περιορισμένος προϋπολογισμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σίγουρα αφήστε που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το Brexit, το οποίο θα μειώσει τον προπολισμό αυτό περαιτέρω. Δεύτερον, όταν λέω ότι τα μάτια μας είναι στραμμένα στο μέλλον, στις μεταφορές ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι και αυτό στραμμένο στο μέλλον. Δηλαδή, δεν έχουμε την πολυτέλεια να εγκρίνουμε προγράμματα που βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά και τα οποία βλάπτουν εν τέλει την οικονομία. Με την έννοια ότι δεν παράγουν, δεν δημιουργούν θέσει εργασία. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σταθμίζει ακριβώ αυτήν την προσθέμενη αξία όταν υπάρχει. Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε υλοποιήσει το α έργο. Και για το Interrail να το συζητήσουμε βεβαίω, πιστεύω ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο, απαραίτητο θα έλεγα εργαλείο. Για δύο λόγου. Πρώτον, πρέπει να προαγάγουμε περαιτέρω την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ε, έργο. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι το διακύβευμα σήμερα. Τώρα, αν αυτό, αυτό το πάσο μπορούμε να προαγάγουμε την διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των νέων, Λέω ναι, ναι, ίσα ίσα πρέπει μάλιστα να το ενισχύσουμε περαιτέρω. Ξέρω ότι κοστίζει 3 δισεκατομμύρια, αλλά τα νιάτα μας νομίζω αξίζουν περισσότερο. Επίσης, είναι κάτι πάλι που μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, ως προς το σου. Πρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω την χρηματοδότηση. Ξέρουμε ότι είναι χρήσιμο, ειδικά το έρασμος. Πλάς. Πώς το βλέπετε αυτό και τέλος. Τα έργα έργα για το μέλλον, το του μέλλοντος. Ναι, φυσικά, συμφωνούμε με όλα αυτά. Μιλήσαμε για τους σιδηροδρόμους. Δεν μιλήσαμε για κάτι άλλο που είναι για μας προτεραιότητα. Δεν μιλήσαμε για την αστική κινητικότητα και την εφορία της. Δεν μιλήσαμε για την ψηφιακή επανάσταση στις μεταφορές. Οπότε το ερώτημα μου είναι προς εμάς, με Y, ε, πώς εσείς βλέπετε τα ζητήματα αυτά και τι ρόλο θα παίξουν στο μέλλον. Ευχαριστώ. να ευχαριστήσω την Πρόεδρο. Πιάνω από εκεί που έκλεισε η Πρόεδρος. Συμφωνώ στις μεταφορές. Χρειαζόμαστε προφανώς μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Πρέπει να ξέρουμε το πλαίσιο. αναφέρεται το Brexit. Τώρα για το 18, το Brexit δεν θα έχει επίπτωση, γιατί το 18 το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχει πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όμως, έχετε απολύτως δίκιο, το πλαίσιο εξελίσσεται, αλλάζει, και αυτό είπε και ο Επίτροπος Έτιγκερ το πρωί. Μιλάμε για δεσμεύσεις 160 δισεκατομμυρίων, ρεκόρ όλων των εποχών, πρέπει να πω. Να μην ξεχνάμε όμως ότι το ποσοστό δεν είναι καθόλου δεδομένο για τα επόμενα χρόνια. Άρα, για το 18 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι στη θέση του. Φυσικά, ναι, καθυστερεί τώρα η έγκριση του νέου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου λόγω Ηνωμένου Βασιλείου και εκλογών. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν και κατά πόσον τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σύγκριση με το 2013. Γιατί έχουμε μια αναθεώρηση μπροστά μα εννοείται. Είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι νέε προτεραιότητες, χωρί καμία αμφιβολία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι και ένα από τους βασικούς ωφελουμένους της αναθεώρηση του ΠΔΠ. Διότι το Horizon 2020 θα έχει μεγαλύτερο προπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη, το κόσμο, το Εράσμος κλπ. Και το Ηνωμένο Βασίλειο θυμίζω είναι ότι είναι μεγαλύτερος ωφελούμενο από το Horizon 2020 γιατί έχει πολύ καλά πανεπιστήμια. Έχει ερευνητικά ιδρύματα υψηλή ποιότητα και κύρου. Όλα αυτά ωφελούνται από το Horizon 2020. Άρα το ξαναλέω, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ωφεληθεί από την αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου που φτάνει μέχρι το 2020. Για το Interrail, επειδή το είπαν πολλοί συνάδελφοι, ήδη έχουμε βασική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής σας και της Επιτροπής των Προπολογισμών. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί Έχουμε εδώ πολλές ε, γνωμοδοτήσεις, είπαν οι συνάδελφοι Βάντεκα, μάλιστα Τέλιτσκα. Όλα αυτά σημαντικά και πρέπει να ξέρουμε αν δαπανίσουμε χρήματα για το Interrail, καταρχάς πώς θα κοστίσει. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα ποσό που είναι αμφίβολο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι τιμή θα δαπανίσουμε για κάθε πολίτη, αν θα υπάρχουν εκπτώσεις και δεν ξέρουμε προς το παρόν τι επιτυχία θα έχει, τι αποδοχή. Δεν ξέρουμε λοιπόν το τελικό κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις στην οικονομία, τις θετικές, δηλαδή οι μετακινήσεις, οι μεταφορές, οι δαπάνες αυτών των ανθρώπων σε διάφορες χώρες, πώς συμβάνουν στις τοπικές οικονομίες κλπ. Εράσμους. Η διεθνή εμπειρία βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των νέων και στην αγορά εργασίας. Ξέρω ότι ένας μήνας ταξιδιού στην Ευρώπη δεν είναι σαν τακτορικό. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα ιδιαίτερα στην ηλικία των 18. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψη της ε, Προέδρου για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Γνωρίζεις νέες χώρες, νέους πολιτισμούς, εξασκείς τις γλώσσες και μαθαίνεις για τα ωφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θέλουμε λοιπόν μια ομαλή εξέλιξη αυτού του προγράμματος ώστε να πάρουμε αποφάσεις και να ξέρουμε και να μάθουμε αν αμφιβολίες που υπάρχουν είναι ουσιαστικές και θα ζητήσουμε πληροφορίες από την Κομισιόν σε συνεργασία εμείς οι δύο επιτροπές και να πιέσουμε την Κομισιόν να μας απαντήσει και να ανταποκριθεί και να ξέρουμε ακριβώς πόσο θα κοστίσει και τι μπορούμε να κάνουμε υπό το τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο και τι στο μέλλον. για το ΕΦΣΥ. Προτείνει κομισιόν του ΕΦΣΥ 2 όπως ξέρετε. Αλλά εγώ έλεγα πάντα ότι το ΕΦΣΥ είναι καλό πρόγραμμα, καλύπτει το κοινό των επενδύσεων, να δούμε όμως ποια είναι η προσταμένη αξία στην καινοτομία, στην ε, συμπληρωματικότητα, στις επενδύσεις. ΕΦΣΥ 2 σημαίνει ότι η εγγύηση από τον προπολογισμό της Ένωσης θα αυξηθεί από τα 16 στα 22 δις. Σε απόλυτους όρους αυτό σημαίνει ότι η συνεισφορά μας θα πάει από τα 8, όχι στα 13, γιατί δεν έχουμε το συντελεστή του 50%. Στα 14 θα πάει για την επόμενη χρονιά για τον προπολογισμό. Η Κομισιόν προτείνει 640 εκατομμύρια. Τώρα το καλό είναι ότι η ΕΚΟΝ και η Μπάτσετ, οι επιτροπές προπολογισμού, είπαν ότι θέλουμε να έχουμε και ένα κονδύλι από το χρηματοοικονομικό εργαλείο του Mobilizing Europe. Αυτό είναι καλό. Να μην ε, έχουμε περικοπές δηλαδή όσον αφορά το εύση για τις δεσμεύσεις. Για τα πιλωτικά τώρα προγράμματα. Συνάδελφοι, η κατάσταση εκεί είναι απλή. Όσοι, μάλλον, όσοι συνάδελφοι υπέβαλαν προτάσεις για αξιολόγηση ήταν οι προτάσεις τους να αποβάλλονται σε αξιολόγηση, ανταποκριθήκαμε δηλαδή. Και πρέπει τώρα να δούμε ποια προγράμματα θα λάβουν βαθμό α ή β από την Κομισιόν. Το ίδιο κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δώσαν προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα και τις προτάσεις που είχαν ΑΒ από την Κομισιόν. Οπότε όσοι συνάδελφοι έχετε υποβάλει προτάσεις με ΑΒ από την Κομισιόν έχετε καλέσει πιθανότητες χρηματοδότησης. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα βελτιώσουμε κάπως και να τα επαναυποβάλουμε ενδεχομένω του χρόνου. Όπως ξέρετε προσπαθούμε να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αλλά η Επιτροπή σας νομίζω όπως και πέρσι θα υποβάλει φέτος ενδιαφέροντα προγράμματα που θα περιληφθούν στο τελικό πακέτο. Aircut. Έχετε δίκιο. Θέλουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν σταθερέ θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες, που θα βασίζονται στην καινοτομία και στην έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι ο ορίζοντας 2020 είναι ένα καλό σημείο κίνησης. Έχουμε και το Connecting Europe, το εργαλείο αυτό. Αλλά όπως είπα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα έχουμε κατανομή των κονδυλίων από το προπολογισμό σε σχέδια και προγράμματα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στους πολιτικούς μας στόχους, αλλά και στην στήριξη τομέων της οικονομίας που οδηγούν στην δημιουργία καλοπληρωμένων και σταθερών θέσεων εργασίας στην κοινοτομία. Σε αρμονία με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε βέβαια. Οπότε εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ευελιξία, υπάρχει ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας για τις επιτροπές τους επόμενους μήνες. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι που με υποδεχτήκατε. Ευχαριστώ για τις πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες που μου υποβάλατε και προσβλέπω στην, στη συνέχεια της συνεργασίας μας τους ε, επόμενους μήνες πριν υιοθετηθεί ο τελικός περιπολογισμός τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον εισηγητή. Είστε πάντοτε ευπρόσδεκτος. Πάντως, μη στεναχωριέστε. Εμείς έτοιμοι είμαστε να σας υποβάλουμε και προτάσεις και παρατηρήσεις για τον προπολογισμό. Και βεβαίως θα το πράξουμε για τον προπολογισμό γιατί δεν θέλουμε επουδενή να μειωθεί ο προπολογισμό μας ως Επιτροπή, αυτό αποκλείεται. Σας προειδοποίησα, έτσι. Ευχαριστώ που ήρθατε και στο επανειδήν. Merci eh. Κύριε Κράμερ, γεια σας, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Κράμερ έχει εδώ μια ομάδα επισκεπτών από το Baden Württemberg, από το Υπουργείο. Σηκώστε το χέρι, εκεί καθέστε. Πολύ ωραία. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλωσορίσατε. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε πάντα συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα των μεταφορών και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις απόψεις σας και σε σας για τα θέματα που εξετάζουμε. Καλώς ήρθατε και πάλι. Συνεχίζουμε με την ημερησιά μας διάταξη. Επόμενο σημείο. εκπομπές σύστημα ανταλλαγών εκπομπών συνεχίση των ισχυόντων περιορισμών το stop the clock όπως λέμε και νομοθεσία που προετοιμάζεται έχουμε τον ε, κανισμό και το άρθρο 55 για το οποίο είχα υποβάλει έτοιμα στην ε, διασκέψη των Προέδρων. Δυστυχώς δεν πέρασε, αλλά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στην κυρία Φώστερ, για να μας παρουσιάσει ακριβώς αυτό το σημείο και το σχέδιο γνωμοδότησης. Κυρία Φώστερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σχολιάσω εδώ για αυτό το θέμα και να πω κάποια πράγματα. Να ευχαριστήσω καταρχάς βέβαια τους εισηγητές και τους συντονιστές, τους σκιώδεις και τους συντονιστές για τη συνεργασία σε σχέση με την ομοδότηση αυτή. Όπως είπατε σωστά, δεν πέρασε το δικό μας και να πω προειδοποιητικά που, ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό θα καταλήξουμε υπό επιτροπή της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και Απασχόλησης. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Και δεν είναι σωστό. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να μας απασχολεί για το μέλλον. Τέλο πάντων, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Ελπίζω οι σκιώδεις να έχουν ένα αντίγραφο της νομοδότησης. Να πω καταρχάς ότι στην εισαγωγή αναφέρω τους λόγους για τους οποίους βρισκόμαστε εδώ σήμερα και να επιθυμίσω στην Επιτροπή μας τους λόγους για τους οποίους καταλήξαμε σε αποτυχία. Επειδή από τους σοσιαλιστές, το ΕΛΚΑ, την ΆΛΔΙΑ, το ΕΣΙΑ, τα μέλη της Επιτροπής μας κατάλαβαν τελικά ότι το ETS για την αεροπλογία δεν είχε κανένα μέλλον, ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, υπήρχαν σοβαρές ε, αντιμαχίες και συγκρούσεις, υπάρχει μεγάλη πίεση όσον αφορά τις εμπορικές ε, συμφωνίες, θέματα παραγγελιών αεροσκαφών και τελικά, σωστά, μαζί με τον Σιμ Κάλλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε όπως αποφάσισε και καθώς το γεγονό ότι ο Επίτροπος μας βοηθάει σε αυτό το θέμα, να πω ότι εμείς είμαστε υπέρ ενό γενικού εγχειρήματο. Εγώ δεν ήθελα βέβαια να το τονίσω αυτό, να είμαστε μη ρεαλιστέ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ένα ευρωπαϊκό τέλο πάντων εργαλείο δεν θα ήταν ρεαλιστικό, γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη απέχηση. Γι' αυτό ακριβώ θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερη δουλειά, θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντά μα σωστά στο Μόντρεαλ και βλέπω ότι τώρα πάνω από 70 χώρες έχουν προσφερθεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κόρσια για τις ανταλλαγές των ρήπων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε. Υπάρχουν και 191 προσυπογράφουσες χώρες στην ε, ΙΚΑΟ μεταξύ των οποίων πολλέ χώρε τη Ένωση, αλλά ως Ένωση εμείς δεν έχουμε, δεν είμαστε συμβλημένο μέλος. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε και τις απόψει των 125 υπολείπων, 165 συγγνώμη, υπολείπων ε, χωρών σε σχέση με το κατά πόσο αυτό το εγχείρημα το Κόρσια θα είναι αποτελεσματικό ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν τα πρωτόκολλα στην ΙΚΑΟ και Πώς λέγαμε, θα πρέπει να εργαστούμε με αυτούς τους περιορισμούς και να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό πάντως προσπαθήσαμε να το καλύψουμε με τροπολογίες και με μια καλή συνεργασία, όπως επίσης και μια καλή συνάντηση που είχαμε στο Μόντρεαλ πέρσι, που ήταν πάρα πολύ παραγωγική και χρήσιμη. Θα δείτε ότι δεν είπα και πολλά όσον αφορά τι τροπολογίε, Συμφωνώ την, με τη θέση τη Κομισιόν, αλλά με κάποιε προσαρμογέ που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Είναι λοιπόν σημαντικό πρέπει οι επιτροπέ στο εσωτερικό τη ΕΚΑΟ να αφηθούν να κάνουν τη δουλειά του. Αυτό είναι σημαντικό και αφορά και τη δικιά μα επιτροπή και την Επιτροπή περιβάλλοντο σε σχέση με το Κόρσια. Εμεί δεν θα πρέπει να γράψουμε, να συντάξουμε το Κόρσια και τι λεπτομέρειέ του. Νομίζω ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ένα τρόπος μέτρησης διεθνής που θα πρέπει να τηρούν και με τον οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται παγκοσμίω. Και μάλιστα ξέρουμε ότι είχαμε και μία πρόβλεψη για τις χώρες του Σέγγεν ως ξεχωριστή οντότητα θα πρέπει λοιπόν όταν έχουμε να κάνουμε τη συμμόρφωση, όταν έχουμε να κάνουμε με τον χαρακτήρα των διεθνών αερομεταφορών, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις πτήσεις ε, εκτός Ένωσης αλλά και εντός Ένωσης. Σε μία λοιπόν από τις τροπολογίες λέμε ότι δεν έχουμε ακριβώς, δεν θα πρέπει να έχουμε μία επικάλυψη σχεδίων σε σχέση με το πώς θα εφαρμόζεται αυτό από τις αεροπορικές εταιρείε, γιατί αυτό δεν θα μας βοηθούσε. Οπότε θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και το αναφέρω μάλιστα, νομίζω στην τροπολογία 3, όπου λέω ότι θα πρέπει τα αντικρουόμενα ή επικαλυπτόμενα σχέδια θα πρέπει να μην θα πρέπει να αποφεύγονται ιδιαίτερα όσον αφορά τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές ε, πτήσεις σε περίπτωση που αποφασίσει με τον τρόπο αυτό μια χώρα μέλος. Θα έπρεπε λοιπόν να αποφύγουμε ένα είδος διοικητικού εφιάλτη, το οποίο θα κοστίσει πάρα πολύ και στην ευρωπαϊκή αεροπλοεία, θα καταλήξουμε σε αντιδικίες όσον αφορά θέματα ανταγωνισμού κλπ. κλπ. Ήθελα λοιπόν να τονίσω εδώ ότι αυτό που κάναμε στην Επιτροπή μας εδώ και που κάναμε καλά, όπως και με τον Γαλιλαίο, για αυτό το πακέτο για τη δέσμη ε, μέτρων και άλλα προγράμματα Clean Sky, Clean Sky 3, Horizon κλπ. Όπως βλέπετε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας ήμασταν πολύ ενεργοί για αυτά τα θέματα και νομίζω ότι αυτό δεν είχε αναγνωριστεί. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το τονίσουμε όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση και μετρίαση των επιπτώσεων των αερομεταφορών. Είχαμε επίσης και τους κατασκευαστές των μικρών αεροσκαφών τους, οποίους είχαμε εξαιρέσει στα πλαίσια του ETS. Είχαμε επίσης εξαιρέσει τις δοκιμαστικές ε, πτήσεις και δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Ε, ξέρω επίσης ότι υπάρχουν ανησυχίε σε περίπτωση που έχουμε εκτροπή αεροσκαφών όταν ξεκινά μια πτήση και τελικά καταλήγει κάπου αλλού για διάφορους λόγους. Τι γίνεται ακριβώς ε, σε αυτήν την περίπτωση, τι ισχύει, μιας και θα έχουμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικά σχήματα ή σχέδια και το Corsia δεν είναι το ίδιο όπως το EU ETS, ή το ευρωπαϊκό δηλαδή ETS. Ε, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Και γι' αυτό ακριβώς διέγραψα κάποια σημεία από το κείμενο της Κομισιόν, γιατί στην Κομισιόν, ε, επειδή έχουμε το άρθρο 28, νομίζω ότι αυτά που θέλουμε να κάνουμε εμείς το καθιστούν περιττό. Και θέλω να πω ότι ένας από τους κύριους τομείς είναι αυτός που αφορά τα μελλοντικά έσοδα. Για το ETS της Ένωσης νομίζω υπήρχε κάποια οριστία. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κλιματική αλλαγή, τις εξελίξεις στον τρίτο κόσμο κτλ. Παρόλο λοιπόν που υπάρχουν προθέσεις καλές, τα χρήματα δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει πάντοτε. Οπότε οποιαδήποτε έσοδα υπάρχουν για, ή υπάρξουν μελλοντικά για τις χώρες της Ένωσης από το ΚΟΣΙΑ, θα πρέπει να επενδυθούν στον τομέα της αεροπλογίας για έρευνα και τεχνολογία ώστε ο τομέας αυτός να στηριχτεί και να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς να κάνει και να δημιουργεί μια καθαρή και πράσινη αεροπλογία, ώστε να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και την πρωτοπορία της αεροπλοείας της Ευρώπης. Κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει αυτή τη στιγμή. Συνολικά πάντως να πω ότι προσπάσα να είμαι απλή εδώ στην γνωμοδότηση και θα έχω και επαφή με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πάντως να πω ότι δεν χάρηκα ιδιαίτερα με κάποια από τα σχόλια, γιατί νομίζω ότι υπήρχε έλλειψη ρεαλισμού για το γεγονό ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε, να επαναυποχωρήσουμε στο ευρωπαϊκό ETS, αλλά αυτό δεν ισχύει αν δεν προχωρήσει το παγκόσμιο σχέδιο. Γιατί το αρχικό ETS της Ευρώπης δεν ήταν αποτελεσματικό και δεν θα είναι αποτελεσματικό για τις τρίτες χώρες αν βρεθούμε σε μια θέση όπου εμείς θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό γιατί θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Και καταλήγω λέγοντας ότι αν εμείς πραγματικά είμαστε σοβαροί για ένα παγκόσμιο σχέδιο η προσέγγιση που έχω και εγώ και οι περισσότεροι συνάδελφοι, τότε αυτό είναι η καλύτερη μας ευκαιρία. Πρέπει να έχουμε μια ενεργητική στάση. Θα πρέπει να σταματήσουμε το ρολόι και να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την υποστήριξη τους σκιώδης και προσβλέπω στα σχόλιά σας ολονών. Νομίζω ότι θα έχουμε και συνάντηση των σκιωδών προσεχώς άμεσα. Αυτά πρόεδρε, που ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φώστερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδης. Ο κύριος Φέρμπερ πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και ζητώ συγγνώμη που έφτασα λίγο καθυστερημένα. Συμμετείχα εκεί στην ε, Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά τα Panama Papers και χρειάστηκε να βρεθώ στη θέση να ε, προστατεύσω τον πρόεδρο της Επιτροπής έτσι, από επιθέσεις εναντίον του προσώπου του. Ε, σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ ε, πολύ για την υποβολή εδώ του ε, σχέδιο γνωμοδότηση. Ε, σε κάθε περίπτωση πραγματικά ευχαριστώ εμφαντικά τη Ζακλίν Φώστερ για το σχέδιο γνωμοδότηση γιατί κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά όλοι μας επιθυμούμε και η αεροπορία να ε, συμβάλλει από τη δική της πλευρά στην μείωση των υπομπών διοξιδίου του άνθρακα. εάν δούμε πώς ιεραρχούνται τα μέτρα εδώ και πού μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τις σχετικέ εκπομπές, τότε τα πιστοποιητικά πραγματικά είναι στην τέταρτη ή στην πέμπτη σειρά, αν θέλετε. Ε, πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να δώσουμε στην καλύτερη διαχείριση της αεροπορίας, δηλαδή νέος ευρωπαϊκός ουρανός και ούτω καθεξής. Μέσω αυτών των μέτρων ήδη έχουν επιτευχθεί 10% μειώσεις των εκπομπών. Δεύτερη προτεραιότητα, υποδομή. Να το πούμε και αυτό εδώ. Για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της ε, Φραγκούρτης ε, δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια ε, ε, μία ακόμα λωρίδα προσγείωσης ε, χωρίς να χρειάζεται πλέον όλα τα αεροπλάνα να κάνουν κύκλους κάθε φορά γύρω από το αεροπλάνο και πίσω να βλέπουμε την ωραία θέα μέχρι να προσγειωθούν. Ε, δηλαδή έχουν γίνει φοβερές εξοικονομήσεις και μειώσεις των εκπομπών ακριβώς επειδή τα αεροπλάνα δεν χρειάζεται να περιμένουν για να προσγειωθούν. Και επίσης νέες τεχνολογίες κινητήρων είναι μια άλλη προτεραιότητα ακριβώς και πάλι με στόχο τη μείωση των εκπομπών. Εάν θέλουμε δηλαδή να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα, φυσικά ε, μοντέρνοι κινητήρες, σύγχρονοι κινητήρες και σύγχρονα αεροσκάφη ε, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκεί δηλαδή ε, μπορούμε να επιτύχουμε και εξοικονομήσει σε κόστο και 5-8% μείωση των εκπομπών. Άρα λοιπόν το πιστοποιητικό εκπομπών ακόμα κι αν λειτουργούσε με τον τρόπο που το είχαμε φανταστεί στην αρχή και δεν θα δημορφωθεί έτσι, ε, μόνο κατά 4% θα συμβάλλει στην ε, μείωση των υπομονών. Οπότε θα θέλαμε να ε, ε, καλέσουμε την ε, κυρία Φώστη να περιλάβει εδώ μία αναφορά ακριβώ στις μεθόδους εκείνες και στους τρόπους εκείνους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο στην μείωση των εκπομπών, πέραν δηλαδή του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Και από εκεί και μετά βέβαια όλο αυτό το σύστημα έχει νόημα εάν υπάρχει και ένας διεθνής συντονισμός. Εάν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να καταστεί παγκόσμιο ζήτημα αυτή η μείωση των εκπομπών, τότε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και παγκόσμια. Δηλαδή δεν θα λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου ε, δημιουργώντας ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι αλλού. Αυτό δημιούργησε ήδη προβλήματα, ένα σύστημα δηλαδή αμυγός ευρωπαϊκό, και τι θα συμβεί ε, αν το συνεχίσουμε. Ε, τα hubs, τα μεγάλα hubs θα δημιουργηθούν στον περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εντός αυτής ε, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αυτό να αποτελεί το στόχο της δική μα στρατηγική. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, έτσι ώστε στον τομέα της έρευνα και τη ανάπτυξη και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που σας ανέφερα, για παράδειγμα μέσω τη επέκταση τη πρωτοβουλία του Ενιαίου μέσω του ΣΥΡΕΝ, να επιτύχουμε ό,τι μπορούμε και σε διεθνέ επίπεδο και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ πως ε, το σύστημα Κόρσια πραγματικά έχει νόημα γιατί ακριβώς εμπεριέχει αυτήν την παγκόσμια διάσταση. Θα πρέπει από εκεί και μετά να αποφύγουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν γιατί και θυμάμαι και τότε όταν είχαμε φτάσει σε ένα συμβασμό μεταξύ ε, Επιτροπής Μεταφορών και Επιτροπής Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS, τελικά οδήγησε στο να πούμε ότι δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο τελικά θα πρέπει να λειτουργεί ε, και παγκοσμίω, αλλά τελικά δεν λειτουργήσε παγκοσμίω. Άρα γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και τώρα θα πρέπει να έχουμε αυτή τη σωστή διεθνή διάσταση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα φτάσουμε εδώ σε ένα καλό κείμενο γνωμοδότησης και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και αποτελεί μια σωστή κίνηση να ε, αναφερθούμε στο πόσο σημαντική είναι η συμβολή της αεροπορίας στη μείωση των εκπομπών, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και ποια είναι η σωστή προτεραιότητα των μέτρων που θα, ληφθούν, που θα πρέπει να ληφθούν σε σχέση ακριβώς με την αποτελεσματικότητά τους για τη μείωση των εκπομπών. Κύριος Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και εμείς ε, θερμά την ε, εισηγήτρια για αυτή την ε, πολύ ε, ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση και εγώ βρέθηκα στο Μοντρεάλ μαζί με άλλους συναδέλφους στο πλαίσιο δηλαδή μιας αποστολής του Κοινοβουλίου και με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής και πράγματι υπήρχε και εκπροσώπηση και από την πλευρά ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι επιχαίρεται πραγματικά το γεγονό ότι δημιουργήθηκαν τα περιθώρια για τη δημιουργία ενό παγκόσμιου συστήματο. Προφανώ ακόμα θα πρέπει να καθοριστούν οι ακριβεί κανόνε, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρείται θετικό το ότι ένα εθελοντικό σύστημα καθίσταται τώρα υποχρεωτικό, ε, ενώ ε, οι περισσότερε, αλλά όχι όλες, οι χώρες είναι διατεθειμένες να προσχωρήσουν σε αυτό. Εγώ είχα διαπιστώσει και στο παρελθόν και εξακολουθεί να ισχύει και τώρα ότι το δικό μας καθήκον είναι να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το παγκόσμιο σύστημα να λειτουργεί εύρυθμα. Δηλαδή όλοι να μπορέσουν να προσχωρήσουν σε αυτό το σύστημα και στην ιδανική περίπτωση ε, ή αν δούμε πραγματικά με θετικό μάτι την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαπιστώσουμε ότι πραγματικά δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα δηλαδή ε, του να υπάρξει ένα τέτοιο διεθνές σύστημα το οποίο θα, μπορέσει, θα είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από όλους. Οπότε τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση η πρόταση της Επιτροπής είναι θετική. Ωστόσο ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η Συμφωνία των Παρισίων να εφαρμοστεί από την πλευρά των κρατών μελών. Τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα σε ό,τι αφορά την κλιματική μα πολιτική. Θεωρώ δηλαδή πω και αυτό αποτελεί ένα πόσπαστο μέρο ε, των προσπαθειών μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, προτάσει που κάνουμε στο πλαίσιο της νομοδότηση τη Επιτροπή Μεταφορών, ε, να πω ότι δεν θα πρέπει να επιδεινώσουμε την πρόταση τη Επιτροπή, θα πρέπει να τη βελτιώσουμε. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Φώστερ και τα όσα περιέλαβε ε, στις δικές της ε, τοπολογίες και ε, νομίζω πως αποτελούν καλή βάση για, την, για τις περαιτέρω συζητήσεις μας. Η εν λόγω συζήτηση βέβαια είναι ενδιαφέρουσα και στο πλαίσιο της Επιτροπής του Περιβάλλοντος, γιατί και εκεί συζητάτε το πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόταση της Επιτροπής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαφάνειας. Είναι σαφές ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία. Ε, εγώ από την πλευρά μου θα υποβάλω τροπολογίε ακριβώ προ αυτή την κατεύθυνση τη διαφάνεια. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Μάση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ πολύ την Τσάκη Φώστερ ε, για, μια, για ένα σχέδιο γνωμοδότηση το οποίο θεωρώ και εγώ ενδιαφέρον. Ε, ε, ο Μάρκο Φέβα ε, ανέφερε πολύ ενδιαφέρουσα πράγματα τα οποία ήθελα και εγώ να αναφέρω και μου έκανε και εντύπωση ότι με κάλυψε τόσα πολλά ε, θέματα. Ε, τώρα, ε, αυτό το αεροσκάφος του μέλλοντος ε, το είχαν ενημερωθεί ε, για το 2011 ότι θα ήταν ένα αεροσκάφος με μηδενικές εκπομπές το οποίο θα είναι κατασκευασμένο πολύ ελαφρύτερα ε, υλικά, ε, το οποίο δεν θα χρησιμοποιείται και τόση ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι έρευνα και καινοτομία είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη βελτίωση της ε, αεροπορίας, γιατί την αεροπορία, τον αεροπορικό κλάδο πάντοτε θα τον χρειαζόμαστε. Οπότε θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις και για την αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη. Από εκεί και μετά. Ο Μάρκος είπε και κάποια πράγματα σε σχέση με την υποδομή. Συμφωνώ, αλλά να πω και εγώ κάτι διαφορετικό. Μία εναλλακτική, αν θέλετε, μια δυνατότητα ε, ε, μέσω της οποίας μπορούμε να επιτύχουμε μείωση των ανθρακούχων εκπομπών ε, στην αεροπορία είναι βελτίωση στα, στους αερολιμένες. Αυτό το taxing, το υπονομαζόμενο δηλαδή, η αναμονή δηλαδή, θα ήταν και αυτό χρήσιμο. Τώρα, ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, το Single European Sky, κατά τη γνώμη μου αυτό η πρωτοβουλία είναι πιο σημαντική. Θα ήθελα κάποια στιγμή επιτέλους να υπάρξει κάποια πρόοδος εδώ. Δηλαδή μόνο ένα δρομολόγιο θα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή για να πάει κανείς, ε, για παράδειγμα, Μπιλπάου ε, ε, για παράδειγμα Φραγκφούρτη, θα πρέπει να κάνει τόσα ζιγ-ζακ ακριβώς επειδή υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το δρομολόγιο που είναι πραγματικά παράλογο. Ε, και πώς μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ε, δημιουργούμε ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών όταν έχουμε επιλύσει τέτοια ζητήματα. Ε, προφανώς είναι θετικό η Επιτροπή να επιτυγχάνει και να είναι ηγέτης σε τέτοια ζητήματα, αλλά διαπιστώσαμε πως στο παρελθόν ότι προσπαθήσαμε ουσιαστικά να επιβάλλουμε σε άλλες χώρες κάτι που δεν επιθυμούσαν. Πράγμα που οδήγησε και στην διακήρυξη της ε, ε Μόσχας, όπου είπαν δηλαδή οι διάφορες χώρες ε, ε, δεν θέλουμε πλέον να διαπραγματεύουμε με την, στην ΙΚΑΟ πλέον αυτό το νέο σύστημα, γιατί οι χαζοί Ευρωπαίοι, εντάξει υπερβάλλω λίγο, έχουν δημιουργήσει το δικό του σύστημα και θέλουν να κάνουν τα δικά τους. εντάξει, η σύμβαση των Παρισιών είναι ήταν μια φοβερή επιτυχία και πραγματικά είναι ιδιαίτερα λυπηρό ο πρόεδρος Τραμπ να προσπαθεί τώρα να ε, την καταστρέψει και πάλι. Ακριβώς για αυτό το λόγο και για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ε, δεσμευτούμε και να ε, επιτύχουμε την, την συνεχιζόμενη διέσμευση ε, με βάση αυτές τις διεθνείς συμφωνίες, ακόμα και αν δεν συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, ίσως καταφέρουμε να τις πιέσουμε τελικά στο να ενταχθούν σε ένα τέτοιο σύστημα, να όλοι οι άλλοι προσχωρήσουμε. Εντάξει, ίσως να είναι ευσεβή πόθη αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά ε, πάντοτε τι προσπάθειε ελάττωση των εκπομπών, θα πρέπει οι προσπάθειέ μα να γίνονται από κοινού. Με όλου δηλαδή, με όλα τα συμβαλόμενα μέρη, όσου ε, υπέγραψαν τη ε, Συμφωνία των Παρισιών. Και ε, επί τη αρχή να πούμε ότι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο ε, έχει ε, υπερψηφίσει και το ψήφισμα της ως στην ε, γνωμοδότηση του Τελίσκα ε, συναδέλφου. Είχαμε εκεί δηλαδή συμφωνήσει με την προσπάθεια που κάνει η ΚΑΟ και το έχουμε λοιπόν ήδη δηλώσει και από εκεί και μετά τονίζω και πάλι την ανάγκη του να προωθήσουμε τις καινοτόμες τεχνολογίες και το πρόγραμμα του Σύμβουλου European Sky. Ευχαριστώ. Καταρχήν για το σχέδιο γνωμοδότησης. Πάντως μιλάμε συνεχώς για το πώς θα σώσουμε τον πλανήτη. Ελπίζω πραγματικά ότι κάποτε θα καταλήξουμε σε μια λύση για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πιστεύω επίσης ότι ο ενίος Ευρωπαϊκός Ουρανός που ανέφερε και Μάισνερ θα μας βοηθήσει να συνεργαστούμε ευρύτερα στους τομείς όπου πρέπει να συνεργαστούμε για να προαγάγουμε την καινοτομία, την μείωση των εκπομπών και τις καλές πρακτικές ανά την Ευρώπη. Αυτό θα μας βοηθήσει όλους. Και θα εξασφαλίσουμε βεβαίως και χρηματοδότηση για κοινά έργα, κάτι το οποίο θα ανακουφίσει και τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα και ο IMO να προτείνει αντίστοιχε λύσεις για τι εκπομπέ στις θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει να βρεθεί μια διεθνής λύση. Αν δεν βρεθεί, τα επόμενα χρόνια, τότε και όλη η ιστορία με τις εκπομπές, τα δικαιώματα κλπ. Όλο το σύστημα αυτό θα στοχίσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλή διαχείριση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Παρακαλώ, λέει πρόεδρος, ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, ζούμε σε έναν κόσμο όπου το κλίμα μεταβάλλεται εξαιτία των εκπομπών, οι οποίε όμω αυξάνονται. Απαράδεκτο. Ιδιαίτερα μετά από το Παρίσι. Η Πράσινη λοιπόν προτείνει το εξή. Από το 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τα μέτρα του το Κόρσια, μέσω του μηχανισμού ETS. 50% όμως των ε, δρόμων πρέπει να εξελιχθούν εκεί που εφαρμόζεται το Κόρσια. Στην αεροπλοεία δεν είναι κίνδυνο μόνο το διοξείδιο του άνθρακα. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, πολλαπλάσιοι μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να αξιολογήσουμε συνολικά τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην μεταβολή του κλίματος, όχι μόνο στις εκπομπές άνθρακα ή διοξιδίου του άνθρακα. Τρίτον, η αεροπλοεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για τις δικές της εκπομπές, όπως έκαναν και άλλοι τομείς. Η αεροπλοεία λοιπόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιθεί είτε να διατηρήσει τις εκπομπές στα ίδια επίπεδα, ούτε πολύ μάλλον βεβαίω να τις αυξήσει. Οπότε, ζητάμε γραμμική μείωση μετά από το 2021. Τέταρτον, στο πλαίσιο του ETS, απαλλαγές πρέπει να δοθούν μόνο σε τομείς όπου υπάρχει κίνδυνος διαφυγής δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει την αεροπορία. Θα πρέπει λοιπόν να επιβληθεί ένα τέλος, ε, ένα, από ένα ευρώ έως πέντε ευρώ σε ευρωπαϊκές πτήσεις. Ε, πιστεύω ότι ακόμα και σε άλλες μεγαλύτερες πτήσεις πάλι η επιβάρυνση θα είναι ελάχιστη. Έτσι θα μπορέσουμε ε, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων. Πρόεδρος, στρέφουμε προς την Επιτροπή. Κύριε Γκράφ, από την Γενική Διεύθυνση κλίματος. Ξέρω ότι το διακύβευμα, όπως λέμε, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια στα θέματα αεροπλοείας, κλίματος και όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει η αεροπλοεία στο κλίμα. Η Κομισιόν, κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω την εισηγητρία για το σχέδιο γνωμοδότηση και τους σκιώδεις βεβαίω εισηγητές για την εν γέννη υποστήριξη της κεντρικής ιδέας της πρότασής μας. Συζητήσαμε βεβαίως σήμερα το πρωί στην Επιτροπή ΕΜΒ τα σχετικά θέματα. Έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση. Να πω λοιπόν δύο λόγια για να θέσουμε ένα πλαίσιο στη συζήτηση. Εμείς στην πρότασή μας ακολουθούμε το τελευταίο ψήφισμα του ΙΚΑΟ για το αγορακεντρικό μέτρο, το Κόρσια, το οποίο είχε ως στόχο να αντισταθμίσει τις εκπομπές θερμολογίας ε, που υπερβαίνουν ενδεχομένω τα επίπεδα του 2020. Ο στόχος μας ήταν λίγο πιο φιλόδοξος, πρέπει να ομολογήσω, όμως ε, ταυτόχρονα η εξέλιξη αυτή είναι καλοδεχούμενη προς τη σωστή κατεύθυνση και αφορά τις εκπομπές της αεροπλοίας σε παγκόσμιο βυσικά επίπεδο. Κάτι το οποίο χρειαζόταν εννοείται. Μετά την COP21, μετά από την συμφωνία που επιτεύχθη στο Παρίσι, τη συμφωνία των Παρισίων, μετά από τη συμφωνία της διεθνούς κοινότητας να προσπαθήσει να περιορίσει την μεταβολή του κλίματος, μάλλον την άνοδο της θερμοκρασίας λόγω της μεταβολής του κλίματος σε κάτω από δύο βαθμούς μετά από τις συμφωνίες να μειώσουμε τις εκπομπές της αεροπλοείας, του τομέα των αερομεταφορών. Ε, όλα αυτά βεβαίως είναι καλές ειδήσει. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά αποτελούν βεβαίως μόνο ένα πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μια λειτουργική εφαρμόσιμη λύση. Η ευθύνη μας είναι να το πετύχουμε αυτό ως το 2021. Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σημαντική από πλευρά πολιτικής, των ψηφισμάτων, των κανόνων που θα θεσπίσουμε. Ο μηχανισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός με άλλα λόγια, όπως είπατε και εσείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον ΕΚΑΟ τρέχουν διαπραγματεύσει όσον αφορά τον χάρτη πορείας, ο οποίος πρέπει να διέπει την εφαρμογή του Κόρσια. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, για παράδειγμα παρακολούθηση, αναφορά, επαλήθευση των εκπομπών, τήρηση μητρών, είναι η ποιότητα των, της αντιστάθμισης κλπ. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτούς τους κανόνες εννοώ. Υπάρχει λοιπόν διαφάνεια και ακρίβεια, ακριβοδίκαιη μέτρηση των εκπομπών. Αυτό θα καθορίσει και την ακεραιότητα και την δικαιοσύνη του επί του συστήματος. Αυτά λοιπόν είναι εξελίξη αυτή τη στιγμή. Οι χώρες που έχουν προσχωρήσει στο Κόρσια εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Και κάτι άλλο που προαναφέρθηκε 67 χώρες πέρσι στη Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΟ δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν τον μηχανισμό, να υιοθετήσουν τον μηχανισμό από την πρώτη μέρα. Αυτή είναι μια πολιτική φυσικά δέσμευση, η οποία τώρα πρέπει να μεταφραστεί σε εθνική νομοθεσία. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει η νομοθεσία, η εθνική νομοθεσία να είναι φυσικά δεσμευτική και αυτό που περιμένουμε να δούμε σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα δεδομένων και κάποιων επιφυλάξεων που κατέθεσαν χώρε. Η Κομισιόν υπεβάλλει τη δική της πρόταση για να διευκολύνει τα περαιτέρω βήματα στον ΙΚΑΟ, τα προσεχή έτη. Έως την επόμενη Γενική Συνέλευση συνεχίζουμε επί περιορισμένου αντικειμένου και αριθμού θεμάτων και μόλις ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά το Κόρσια, όταν ε, ξεκαθαριστούν οι κανόνες δηλαδή και δούμε τι έχει κάνει κάθε χώρα, τότε θα προβούμε σε μια διαμεσή αξιολόγηση. Αυτό είναι η πρόταση της Κομισιόν. Με δύο λόγια. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανάγκη να υιοθετήσουμε τάχιστα την πρόταση αυτή διότι αν δεν ε, την εγκρίνουμε ε, γρήγορα, τάχιστα, δηλαδή ε, στα τέλη του έτους του 2017 και σίγουρα πριν την έναρξη του νέου κύκλου συμμορφής, τότε ξαναγυρνάμε στην αρχή και δεν θέλουμε φυσικά να προκαλέσουμε αναταραχή μεταξύ των εταίρων μας, ούτε να θέσουμε υποαφισβήτηση τα όσα έχουμε επιτύχει ως σήμερα στον ΙΚΑΟ. Υπό την ενία αυτή, εμείς από την πλευρά τη Κομισιόν θα διευκολύνουμε την επίτευξη σύμφωνη μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τι τρέχουσε εξαιρέσει και την διαμεσή αναθεώρηση, η ευθύνη μα είναι, εννοείται, να δώσουμε χώρο και χρόνο στον ΙΚΑΟ να προτείνει συγκεκριμένου ρεαλιστικού εφαρμόσιμου κανόνε και να προετοιμαστεί φυσικά για την αναθεώρηση. Η αναθεώρηση και η αξιολόγηση θα αφορά τις εξελίξεις τους στόχους που έχουμε θέσει το 2030 και συνεχώς περιμένουμε και η αεροπλοία να συμμετάσχει στην προσπάθεια με βάση τους στόχους του 2020. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Η πρότασή μα θα ήθελα να πω, είναι ουδέτερη. Έχουμε μπροστά μα κάποιε εναλλακτικέ λύσεις, αλλά δεν θέλω να προδικάσω καμία εξέλιξη στη φάση αυτή, γνωρίζοντα βεβαίω ότι πρέπει να αποφύγουμε και επικαλύψει στο έργο μας. Όπω είπε η κυρία Φώστερ, το Κόρσια αφορά αντιστάθμιση. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα για αντισταθμιση ενώ το ETS αφορά την παραγωγή στις χώρες μέλη. Πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ σημαντική διαφορά εν ώψη του 2030 και των στόχων που έχουμε θέσει για το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα μέτρα, τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε και άλλο. Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμαστε το Κόρσια, και το ETS. Το ETS για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να βεβαιωθούμε το σύστημα των δυνατών ότι το σύστημα λειτουργεί, αποδίδει, αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι αποδίδει πολλά. Κάθε χρόνο. Είναι Ε, Δύο ακόμη παρατηρήσεις για το Κόρσια. Το υποστηρίζουμε φυσικά, θέρμος, το υποστηρίζουμε, αλλά και εδώ, προσοχή. Να μην δώσουμε την εντύπωση ότι είναι το τέλειο εργαλείο. Γιατί με το πρόβλημα των εκπομπών τη Όχι. Ο μηχανισμός εξελίσσεται. Δεν έχει ακόμη φτάσει στο, στην τελική του μορφή. πάντως έτσι δείχνουμε ότι είμαστε προσιλωμένοι στον στόχο, τον παγκόσμιο στόχο της αντιμετώπισης της μεταβολής του κλίματος. Θα συγκεράσουμε τις δισταμένες ανάγκες. Τώρα, όπως ε, είδατε και στην πρότασή μας, έχουμε περιλάβει και μία αναφορά στον παράγοντα γραμμικής μείωσης μετά από το 2020 στο πλαίσιο του ETS, εάν συνεχίσουμε φυσικά και με την επιφύλαξη της αναθεώρησης και αξιολόγησης. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν για να είμαστε στο ίδιο μήκος κειμένου με τους άλλους τομείς που συμμετέχουν στο ETS. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση συνέχεια και συνέπεια μετά τους στόχους που θέσαμε το 2013. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά λίγο πολύ. Θα είμαστε εννοείται σε επικοινωνία, θα τα δούμε αυτά και με την αφορμή, με αφορμή τις τοπολογίες που θα καταθέσετε. Από εδώ και πέρα εμείς θα συνεργαστούμε στενά μαζί με όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκράφ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Γρήγορα θα δώσω το λόγο για πάση κυρία Φώστα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τους αναλογούς και την Κομισιόν η Κομισιόν είπε τον γραμμικό συντελεστή κάτι σχετικά με αυτό και την αρχική αναφορά στο πρώτο έγγραφο και τροποποίηση. Είναι δύσκολο να θεσπίσουμε ένα γραμμικό συντελεστή τη στιγμή που να κάνουμε τελείω διαφορετικό σχέδιο και γι' αυτό ακριβώ το λόγο το αφαιρέσαμε. Τελείω διαφορετικό μέτρο δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή η συνετή προσέγγιση της Κομισιόν. Είτε συμμετέχουμε είτε δεν συμμετέχουμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνουμε συζητήσεις στο Μόντρεαλ. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλή συμφωνία πάντως. Τώρα για τους συναδέλφους να πω για τον Μάρκος Φέμπερ ότι σωστά μιλάει Νομίζω ότι δεν πιέζονται αρκετά οι χώρες μέλη. Ξέρουμε ότι έχουμε δυνατότητες στα αεροδρόμια, ξέρουμε ότι έχουμε ε, προβλήματα στις διάφορες χώρες ε, με αιτήσει ε, όσον αφορά επεκτάσεις αεροδρομίων, αεροσκάφη, καύσιμα κτλ. Ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν είναι καλά για το περιβάλλον, αλλά ούτε και για τους καταναλωτές. Οπότε θεωρούμε ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν τις ευθύνες τους. Και κάτι άλλο υπόθηκε για τον νέο ευρωπαϊκό χώρο, ε, νέο ευρωπαϊκό ουρανό δηλαδή, παρόλο που υπάρχουν κάποια ζητήματα με την εφαρμογή, δεν υπάρχουν ζητήματα με, την νέο, με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, και θα πρέπει και πάλι να υπάρξει η απαραίτητη βούληση και οι χώρες μαλλί θα πρέπει να τηρήσουν την νομοθεσία και τους κανονισμούς που υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Ο κ. Νίλς αναφέρθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού και πρέπει να πω ότι συμφωνώ. Δεν περιλαμβάνονται αεροπλοεία και ναυσιπλοεία στην Συμφωνία του Παρισιού. Αλλά ίσως αυτό να είναι και πλεονέκτημα. Ίσως επειδή δεν αναφέρονται επειδή οι Αμερικανοί δεν ξέρουν ακόμα θέλει να κάνει ο Τραμπ αλλά ίσως να μην θέλει να σε μετάσχει στην Συμφωνία του Παρισιού. Αν λοιπόν οι Αμερικανοί κάνουν κάτι τέτοιο, δεν τους αποτρέπει αυτό να προσχωρήσουν στο Κόρσια. Οπότε αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε δεν νομίζω ότι τους αποτρέπει από το να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Κόρσια. Και εγώ μίλησα με διάφορους συναδέλφους από την Αμερική. Κάποιες χώρες και είπα, νομίζω ότι το εξετάζουν σοβαρά, γιατί νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων τελικά. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτό θα εκτυλιχθεί σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Η κυρία Κίλεναν, η καλή μου φίλη, επίσης μίλησε για την τεχνολογία το Clean Sky και το καινούριο Clean Sky 3 που έρχεται. Εμείς θα πρέπει να συνεχίζουμε να ηγούμαστε σε αυτό τον τομέα και να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε γύρω από τα αεροδρόμια όπου έχουμε συμφόρηση να είναι ευθύνη της χώρας ε, μέλου ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα αεροδρομία και χρησιμοποιούμε την βέλτιστη τεχνολογία και τα βέλτιστα συστήματα για να μειώσουμε ακριβώς την ρήπανση και τις εκπομπές από όλες τις μορφές μεταφορών. Όχι μόνο από το τμήμα Σας είπα τις παρατηρήσεις μου για τα σχόλια των σανδέλφων. Θα έχουμε και επαφές με τους σκιώδεις και θα πρέπει νομίζω να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και με άλλους ενδιαφερόμενους από άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, αλλά συμφωνώ ότι έχουμε και ένα χρονικό περιορισμό και θα ζητούσα από τους αδελφούς να εξετάσουν σοβαρά το τι θα καταθέσουμε ως τροπολογίες, γιατί όσο πιο λίγο, όσο λιγότερο επίμαχο, τόσο το καλύτερο. Θα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν το ρολόι και θα πρέπει, έστω και αν έχουμε αποκλίνουσε απόψει να ομονοήσουμε σχέση με το πώ θα λειτουργεί το νέο σχέδιο. Νομίζω ότι η προτεραιότητα, ξαναλέω, είναι το να σταματήσουμε το ρολόι, να σταματήσουμε το χρόνο. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πρόεδρε και προσβλέπω βέβαια τι συναντήσει με του ανδρού για να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριε Φώστερ, να υπενθυμίσω ότι οι προθεσμοί για την κατάθεση τροπολογιών είναι 6 του Ιούνιου το μεσημέρι, 12. Αυτά. Πάμε σε ένα άλλο καυτό θέμα. Για τις εσωτερικές οδούς, πλουτές οδούς και μεταφορές. Έχετε εδώ την υποφαινόμενη που είναι και εισηγήτρια για αυτό το θέμα. Μη φύγετε, μη φύγετε, θα είναι ενδιαφέρον. Euh, Πάμε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Κατάργηση του κανονισμού 11.01.89 του Συμβουλίου και των κανονισμών 28.88.2000 και 6.85.2001 του Συμβουλίου. Είχαμε το ρηφί της ε, Κομισιόν για καλύτερο νομοθεσία, τη βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να παράσχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της, ενδιάμεση... της διοργανικής συμφωνίας συγγνώμη, μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου Κομισιών για την ενίσχυση της διαδικασία νομοθέτησης και κατάργησης των παρεχημένων νομοθετικών εργαλείων. Καταρχάς, το 11.01 όσον αφορά την, ε, τις πλωτές εσωτερικές οδούς, στην Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία. Στόχος λοιπόν εδώ είναι να μειωθεί ή να υποχωρήσει τέλο πάντων το υπερβάλλον δυναμικό ώστε να υπάρχει ένα συντονισμό με τη χωρητικότητα αυτών των σκαφών σε κοινοτικό επίπεδο. Ο 7-18 τώρα το 89 του Συμβουλίου Αφορά και αυτό στις εντορικές πλωτές οδούς και την πρόθεση των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών εδών τροποποιήθηκε ώστε να συνεχίσει να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία ο τομέας της ε, να ιδιαίτερα όσον αφορά το δυναμικό και Έχουμε τον 1101 του 89 επίσης, που και αυτός είναι παροχημένος και ο οποίος θα πρέπει και αυτός να καταργηθεί. Μιλάμε επίσης για τον 2888 που κάνει την κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων χωρομελών όσον αφορά τις μεταφορές με την Ελβετία από το 2001 μέχρι το 2004 μεταφορά και εμπορμάτων αλλά και επιβατών σιδηροδρομικά και οδικά από την 1η πρώτου του 2005 ίσχυε αυτός ο κανονισμός, δηλαδή είχαμε μέγιστο βάρος 40 τόνους και δεν είχαμε υποχρέωση για αδειοδότηση και άλλους περιορισμούς. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο κανονισμός είναι παροχημένος και θα πρέπει να καταργηθεί και αυτός και τέλος. Ο 685 κανονισμός. Με παρακολουθείτε όλοι, σας βλέπω λίγο χαμένους. 685 λοιπόν 2001 που καθορίζει τους κανόνες κατανομής, η δικλίδα κατανομής, μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Δημοκρατίας Βουλγαρίας και μεταξύ Ρουμανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικός και την πρόθεση των συνδυασμένων μεταφορών. Παρχημένος και αυτός, επειδή η Βουλγαρία βέβαια και η Ρουμανία επίσης προσχώρησαν στην Ένωση Οπότε ως χώρες μέλη βεβαίω, δεν υπόκεινται λογικά σε κανένα καθεστώς αντιδότησης όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, παροχημένος και αυτός και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να καταρριχθεί πρώτα. Σας το πάω λίγο γρήγορα να δω αν είσαστε ξύπνοι, λέει η Πρόεδρος, για αν κοιμηθήκατε. Προτείνω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να αποδεχτούμε την κατάργηση αυτών των διαφόρων κανονισμών. Θέλετε να σας δώσω και τα στοιχεία. Έτσι, μη σας πω τώρα τα στοιχεία, θα κάνουμε πάρτι. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο και τις χώρες μέλη που πρότεινα να υιοθετήσουμε, μάλλον πρότεινα να υιοθετήσουμε την πρόταση της Κομισιόν, κάνοντας όμως κάποιες τροποθετήσεις, τροποποιήσεις στα εκτιμώντας και συγκεκριμένα έχουμε δύο αλλαγές μετά από δικό μας αίτημα. Και ελπίζουμε όλα αυτά να περάσουν στην πρώτη ανάγνωση. Χωρίς τροπολογίες. Ώστε να αποφύγουμε τους μακροσκελείς και δύσκολους τριμερείς διαλόγους που καμιά φορά είναι δύσκολοι. Τώρα, η Κομισιόν. Ποιος εκπροσωπείται την Κομισιόν. Γεια σας, γεια σας, καλά είσαστε. Πώς πάει, λέει ο Πρόεδρος. Η Κομισιόν λοιπόν που λέγαμε να μας απαντήσει για το εξής. Εδώ και καιρό είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι κανονισμοί που αναφέραμε έχουν καταστεί παροχημένοι, θα πρέπει να καταργηθούν κτλ. Ερώτημα. Εύλογο. Γιατί περιμένατε τόσο καιρό για να μας κάνετε προτάσεις, γιατί χάσαμε πολύ καιρό, λέει η Πρόεδρος. Αλλά πριν σας δώσω το λόγο, να μιλήσουν πρώτα συνάδελφοι. Κυρία Μπίν, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σκεγγραφίσατε σωστά το περιεχόμενο των κανονισμών που είναι παροχημένοι. Δεν θα επαναλάβω τους λόγους για τους οποίους είναι παροχημένοι. Είναι καλό που κάνουμε έτσι ένα σημάζεμα και στο refit της Κομισιόν και που απλουστεύουμε και βελτιώνουμε την νομοθεσία. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπατε και συμφωνώ με τις δύο τροπολογίες που προτείνατε. Και ελπίζω όπως και εσείς να περάσουν όλα αυτά στην πρώτη ανάγνωση για να αποφύγουμε τους τριμερούς διαλόγους. Ευχαριστώ λοιπόν για την ε, παρουσία σας Πρόεδρε και θέλω να πω ότι την αποδέχομαι απολύτως και τη στηρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κλίν. Ο κύριος Ρικέ, όχι, δεν θέλετε. Euh, Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Λέει ο κύριο Ρικέ. Ιδιαίτερα συμφωνώ με τι δύο τροπολογίε που θα μα επιτρέψουν να παρακάμψουμε τον τριμερή διάλογο και τη δικασία στην αλλαγή. Κύριε Μέστινα, έχετε λόγο καθώς ο αντιπρόεδρος ε, ε, της, ε, εδώ της Επιτροπής μας που εκπροσωπεί και την πολιτική μας ομάδα ήδη συμφώνησε, δεν έχω πολλά να πω. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τη διαδικασία που προτείνατε εσείς κυρία Πρόεδρος Συγκήτρια. Ευχαριστώ. Ωραία. Βλέπετε να επιτροπή ότι είμαστε εδώ ομονοούντες, ομόφωνοι. Οπότε Κομισιόν πρέπει ούτως να απαντήσετε στο αρχικό μου ερώτημα. Η κυρία Βέρνερ, ε, πώς σας λέμε Βέρνερ. Βέρνερ. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε τις νέες προτάσεις, τις νέες προσπάθειες, συγγνώμη, της Επιτροπής ε, Juncker για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασία ώστε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια και σαφήνεια. Γι' αυτό εδώ και τρία χρόνια ε, εξετάζουμε τον μακροσκελή κατάλογο του κεκτημένου των μεταφορών για να δούμε ακριβώς ποια νομοθεσία είναι πια περίτη ή παροχημένη όπως αυτές που αναφέρατε σήμερα για τις οποίες χρειάζεται μια πράξη κατάργησης. Είναι λοιπόν παροχημένες αυτές οι αποφάσεις και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Με αυτές τις αποφάσεις δηλαδή. Πρόσφατα είδατε και στο σιδηροδρομικό πακέτο αλλά και για τις εσωτερικές πλουτός οδούς ότι καταργούσαμε παλαιότερες νομοθετικές πράξεις ταυτόχρονα όμως με την υποβολή νέων προτάσεων. Εδώ έχουμε ακόμα δύο προτάσεις πάνω στις οποίες δουλεύουμε και που είχαμε ανακοινώσει στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας μας ε, για το 2017. Αν θέλετε να σας δώσω τους αριθμούς, αλλά και πάλι πρέπει να σας υποβάλουμε συγκεκριμένη πρόταση για κατάργηση, που ελπίζω να λάβετε σύντομα. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε και να ερευνάμε προσεκτικά το κεκτημένο κάθε φορά που βάλουμε πρόγραμμα εργασίας. Αν βρούμε και άλλα νομοθετικά στοιχεία παροχημένα, δεν θα διστάσουμε να υποβάλουμε νέες προτάσεις. Με στόχο να έχουμε ένα κεκτημένο όσο πιο επίκαιρο γίνεται. Αυτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κυρία μου, λέει η Πρόεδρος. Αν έχετε και εμπνεύση, μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι τις 7 του Ιούνιου στις 2 το απόγευμα. Αν δεν έχετε έμπνευση, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, λέει ο Πρόεδρος. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες τροπολογίες. Θα έχουμε τώρα μια συνάντηση συνεδρίαση μάλλον και κλεισμένων των θυρών. Οπότε επειδή θα συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών, θα παρακαλέσω από τους μη, μη έχοντες εργασία να αποχωρήσουν. Βέβαια, όλα τα μέλη, βουλευτές και το προσωπικό τους μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα. Αναμένουμε λοιπόν την αποχώρηση.